Λοιπόν, πάμε στην ημερήσια διάταξή μα. Έχουμε στάσει των συντονιστών της συνεδριάς 24 Σεπτεμβρίου. Απεστάλησαν τα κείμενα ηλεκτρονικά. Δεν έχω λάβει κάποιες παρατηρήσεις. Άρα είναι εγκεκριμένα τα κείμενα. Πάμε στις ψηφοφορίες. Σας παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες για την ψηφοφορία, διότι θα έχουμε από την αρχή κάποιες ψηφοφορίες που θα υπάρχει μικρή διαφορά ψήφων. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη γνωμοδότηση ΚΑΟΤ που αφορά το άρθρο 106 Ξεκινά λοιπόν η ψηφοφορία. Την ένσταση λοιπόν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Μπορούμε να τελειώσουμε την ψηφοφορία. απορρίπτεται με 34 ψήφους κατά, 30 υπέρ και 3 αποχές. Πάμε λοιπόν σύμφωνα το άρθρο 106 στην άλλη ένσταση για τον κανονισμό που αντικαθιστά το παράτημα 3 της οδηγίας 98-2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ανάκριση κάποιων οδηγιών. Η κυρία Κώστινγκέρ συνέταξε, έκανε την πρόταση. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται με 39 Ψηφού 21 ε, υπέρ και 7 ε, αποχές. Πάμε στο σημείο 12 και σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένσταση τη συνάδελφου Κέστιγκερ βάσει του άρθρου 106. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 40 ψήφια εναντίον, 20 υπέρ και 7 αποχές. Andiamo al punto 13. Σημείο 13. διαπραγματευτική εντολή για την οδηγία που αφορά τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται να ψηφίσουμε για τις πλαστικές σακούλες. Ήταν πολύ ισχυρή ψηφοφορία στην προηγούμενη θητεία με καλή συμβαστική λύση. Υποστήριξαν όλες οι ομάδες εκτός το ECR τότε και βάσει της πρώτης ανάγνωσης ζητώ την υποστήριξή σας για να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεων το Συμβούλιο. Χρειάζω λοιπόν να μου δώσετε την εντολή για να μπορέσουμε να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία για την εντολή χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία. Το ΕΛΚ αυτή τη στιγμή έχει έναν ψηφοφορό παραπάνω. Κάποιον, α, κάποιον απληρωματικό μέλος του ΕΛΚΑΝ έχει την καλοσύνη να αποσύρει την κάρτα. Πέρα ψηφοφορίας. Εξήντα οκτώ ψήφι υπέρ. voto più forte di così, collega Καλύτερα από έτσι δεν μπορούσε να πάει η ψηφοφορία, συνάδελφε Όκεν. Λοιπόν, η αντιπροσωπεία που θα πάει στον τριμερή διάλογο για τις συνομιλίες θα παρτίζεται από την κυρία Άουκεν, από την υποφαινόμενο σαν πρόεδρο της Επιτροπής, συνάδελφο Οβενή του ΕΛΚ, Μποναφέ για τους σοσιαλιστές, Γκέρλινγκ για το ECR, Γκέρμπεντι για την Άλτε, Φορένσα για την ΚΟΕ και Εύη για το FTT. Σημείο 14. Stiamo cercando il collega Favia. Ε, ε, Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή για να αναφερθεί στο σημείο αυτό. Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε, όπως και οι συνάδελφους, η κυρία Άουκεν, και εγώ ήθελα να ζητήσω την ψήφο σας για την παρακολούθηση αυτή για τις ε, άνθρακα και θαλάσσιες μεταφορές, για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και περιμένω την ψηφοφορία. Χρειάζεται απόλυτη ψηφοφορία. Ξεκινά η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. 59 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά και τρεις αποχές. Η διαπραγματευτική ομάδα, πέρα από τον συνάδελφο Φαρία, θα παρτίζεται από τον πρόεδρο, τον υποφανόμενο, κύριο Φιέλνερ για το ΕΛΚ, Γκούτλαντ για τους σοσιαλιστές. Δεν έχουμε από το ECR κάποιο όνομα. Ο συνάδελφος Duncan λοιπόν για το ECR. Abounds για την Good, Λόβιν για τους πράσινους και Flont για το FTT. Και τώρα, στο επόμενο σημείο, το 15, εν ώψη της διασκέψεως COP20 στη Λίμα. Έχουμε προφορική ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. για τη συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών το 2014 Βλέπετε, έχετε όλη την προφορική ερώτηση. Μπορούμε δυνατά σας χειρός να ψηφίσουμε. Είναι εύκολο αυτό. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η δεύτερη προφορική ερώτηση για το Συμβούλιο και αυτή πρέπει να εγκριθεί δυνατά σας ισχυρός υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Στο επόμενο σημείο, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για την οικονομική πολιτική, η υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2014, η συγητής για την γνωμοδότηση ήταν ο συνάδελφος Γκερμπράντι. Αν θέλει μπορεί να δώσω το λόγο ή μπορούμε να ψηφίσουμε άμεσα. Μπορούμε να ψηφίσουμε αμέσως. Ξεκινάμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. σα στις χειρός ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά. Ας κάνουμε μια παλήθευση ηλεκτρονική. Ψηφίσατε όλοι. Μπορεί να κλείσει η ψηφοφορία. απορρίπτεται. 36 κατά 32 υπέρ, καμία αποχή. Τροπολογία 2 που είναι συμβατή με την 1. Ο εισηγητής είναι κατά, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι είναι παρόμοια ισορροπία, αλλά κάνουμε μια παλήθευση να είμαστε σίγουροι. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 34 ψήφοι κατά, 31 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 3 της συναδέλφου Κονέτσνα υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι είναι η ίδια ισορροπία όπως πριν. Άρα απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ιβασκίεβιτς. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Μέλο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 κονέτσνα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 1 πέντε πολιτικών ομάδων υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Πέντε πολιτικών ομάδων υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ιβασκεβιτς Υπέρ. Κανείς υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Γκέρλινγκ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Πέντε πολιτικών ομάδων υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Κονέτσνα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. απορρίπτεται. Έκανα λάθος λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 13. Γραμματικάκης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Κερμπράντι. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Γκέρλινγκ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Μέλο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Σκλέκ. Καταπίπτει. Τροπολογία 18. Συμβατή με τις άστροπολογίες. Γραμματικάκης υπέρ. Οι τροπολογίες 15 και 16 έχουν απορριφθεί, άρα ψηφίζουμε τροπολογία 17. Σκλεκ υπέρ της 17. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19 κονέτσνα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 Γκέρλινγκ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Γκέρλινγκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Σκρλέκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23, Γκερμπράντι, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24, Σκελέκ, υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. πολύ ισορροπημένη η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 25. Τροπολογία 26. Γκέρλινγκ. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 πεντιτσίνη σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 28 σκρλέκ υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Τροπολογία 29, σκρλέκ, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 30, σκρλέκ, υπέρ, κατά, άποχες έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 37 ψήφι κατά τροπολογία 31 καπούτο υπέρ κατά Αποχές. Και εδώ θα κάνουμε έναν έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Όλες οι άλλες τροπολογίες Οι 32 και οι 33 καταπίπτουν. Έχουμε τη συμβαστική 4. Υπέρ τη συμβαστική 4. Κατά άποχες εγκρίνεται. Οι άλλες τροπολογίες καταπίπτουν. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία κάνουμε την τελική μας ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν με 53 ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή. Πάμε στο σημείο 17. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Πάμε στο σημείο 17. θα μιλήσουμε για τη διάσκεψη της Λίμα για την αλλαγή του κλίματος. Κατάλαβα ότι τελειώσαμε την ψηφοφορία, αλλά αυτός που ενδιαφέρεται να παραμείνει, ας παραμείνει κάνοντας ησυχία, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες. Όποιος επιθυμεί να εγκαταλείψει την αισθούσα ας το κάνει ήσυχα, παρακαλώ, ούτως ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες της Επιτροπής. Σαν εισηγητής θα προβώ σε μια σύντομη εισαγωγή όσον αφορά την πρόταση ψηφίσματος που έχουμε ετοιμάσει. Και μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους θα προβούμε σε παρεμβάσεις. Θα γίνει ένας γύρος ανταλλαγής απόψεων. Σε αυτή την πρόταση ψηφίσματο συνοψίζουμε κάποιες σημαντικές πτυχές που παραδοσιακά στηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της διεθνούς συζητήσεως για την κλιματική αλλαγή το σχέδιο ψηφίσματος παρουσιάζει μια έποψη πιο φιλόδοξη εν ώψη της τελικής διατύπωσης της θέσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την διάσκεψη COP20 θα γίνει στη Λίμα. Χρειάζεται κατεπηγόντως δράση. Θα πρέπει όλα τα κράτη να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές τους των αερίων του θερμοκηπίου. Τέτοιες εκπομπές Σύμφωνα με το διακυβερνητικό πάνελ για την κλιματική αλλαγή, θα έπρεπε να φτάσουν πολύ σύντομα στη μέγιστη ακμή και μετά να μειωθούν τουλάχιστον κατά 50% μέχρι το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 ούτως ώστε να παραμείνει μια λογική πιθανότητα η αύξηση της θερμοκρασίας, μέση θερμοκρασία στον κόσμο να, παραμείνει κάτω από τους δύο βαθμούς σε σχέση με την πρώτη βιομηχανικής περίοδου εποχής. Μια πρόοδος προς τη συμφωνία το 2015. Η διάσκεψη της Λίμα θα πρέπει να θέσει επιτάπητο τα βασικά στοιχεία της Διεθνούς Συμφωνίας που προβλέπεται για το 2015 βάση προόδου που θα έχει επιτευχθεί το 2014 στα πλαίσια της πλατφόρμας του Durban. Θα πρέπει να τονίσουμε ποιε είναι οι φιλοδοξίε μα. Αυτό το κάνουμε στην πρόταση πριν το 2020 ποιε είναι οι φιλοδοξίε. Όλα τα μέρη θα πρέπει να προβούν σε μια πολυμερή αξιολόγηση τη επιτευχθή σα προόδου σχετικά με τους στόχους της μείωσης των εκπομπών για το 2020 για να εξαλειφθεί τη τεράστια διαφορά που υπάρχει μεταξύ επιστημονικών στοιχείων και των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα διάφορα συμβαλόμενα μέρη θα πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται όσον αφορά τη χρηματοδότηση το κλίμα. Όλα τα μέρη θα πρέπει να συμβάλλουν σύμφωνα την ποσόστοσή του στι δεσμεύσει που ανέλαβαν σύμφωνα με τη Συμφωνία τη Κοπενχάγη για να κινητοποιηθούν από κοινού 100 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο μέχρι το 2020. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτή θα πρέπει να αυξήσουν την κινητοποίησή των πόρων του για το κλίμα και στο τέλος ε, προσθέσαμε κάποιες πτυχές όσον αφορά ε, τις, ε, τις θαλάσσιες μεταφορές, ξαρομεταφορές, φιλόδοξοι στόχοι για να πετύχουμε και σε αυτούς τους τομείς ικανοποιητικά αποτελέσματα εγκαίρως και στα πλαίσια της ΙΚΑΚ και του IMO για τη μείωση των εκπομπών των αερίου του θερμοκηπίου στις θαλάσσιες και ενέργειες μεταφορές μετά από αυτή την σύντομη παρουσίαση όσον αφορά το περιεχόμενο και το ψήφισμα θα ήθελα να ξεκινήσουμε το γύρο ανταλλαγής απόψεων. Ας ξεκινήσουμε από το ΕΛΚ. Ε, ο συνάδελφος Μπέλετ έχει το λόγο. Ε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στη Νέα Υόρκη, εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να δηλώσουμε ότι είμαστε βαθιά προσιλωμένοι σε αυτή την προσπάθεια με φιλοδοξία, υποστηρίζουμε τον ΟΗΕ, όπως είπατε Πρόεδρε, και θέλουμε να είναι και δεσμευτικά, νομικό, δεσμευτικό, νομικά δεσμευτικό, Ε, στη Λίμα προετοιμάζεται η σύνοδος του Παρισίου. Έχουμε πρόβλημα με τη μετάφραση. Σε ποια γλώσσα. Okay. you the problem? Okay. Εντάξει, με τα ακουστικά ήταν μάλλον. Ωραία, ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ανακεφαλαιώνω και ζητώ συγγνώμη. Ε, είναι δικαιολογημένος από όνο Κάχαρης Φλόρενς γιατί σε άλλη συνεδρίαση. Τι πρέπει να κάνουμε, δύο-τρία σημεία. Ε, βεβαίως θα πρέπει να έχουμε όλη την ίδια φωνή και στο Παρίσι και στη Λίμα και η Σύνοδος Κορυφής τέλη Οκτωβρίου 23 και 24 ε, θα είναι μια κρίσιμη επόμενη φάση. Θα πρέπει να ζητήσουμε μια σαφή ε, δέσμευση και πάλι από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ότι είμαστε προσελωμένοι σε αυτό το στόχο η υπερθέρμανση ε, του πλανήτη να περιοριστεί κάτω από δύο βαθμούς Κελσίου. Επίσης θα πρέπει να είμαστε σαφείς στο INDC, στην πληροφόρηση ε, εκ των προτέρων που δίνουν οι χώρες, οι συνεισφορές των κρατών δηλαδή να είναι δεδομένες και συγκρίσιμες προφανώς και να υπάρχει και μια σαφήνεια σε ό,τι αφορά την εκ των προτέρων λοιπόν ενημέρωση έτσι ώστε και στη Λίμα και στο Παρίσι να γίνει δυνατή μια συμφωνία που να βασίζεται σε κοινά συγκρίσιμα ε, στοιχεία. MRV το επόμενο θέμα που είναι η παρακολούθηση, η αναφορά και η επαλήθευση στα αγγλικά τα αρχικά. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει πάρα πολύ καλή και αξιόπιστη ε, ρύθμιση για αυτά και υποχρεωτικά ε, να έχουμε ελέγχους και αντίβαρα μηχανισμούς ε, συμμόρφωσης, μηχανισμούς ελέγχουν όλων αυτών των προσπαθειών που γίνονται. Θα πρέπει να τα κάνουν αυτά και τα κρατη και οι υπογράφοντες της ε, ε, τερχόμενης συμφωνίας. Δεν είναι λοιπόν μόνο η συμφωνία, αλλά πώς εφαρμόζεται και πώς ελέγχεται η εφαρμογή της. Και ένα τελευταίο πρόεδρο που θέλω να πω είναι ε, ένας βιώσιμος, σταθερός και διαρκής μηχανισμός για την τιμολόγηση του διοξιδίου του άνθρακα. ο Γενικός Γραμματέας του Ιεμπάν Κιμούν ε, εκφώνησε ένα λόγο στη Νέα Υόρκη και τα διατράνωσε και αυτά και πάλι. Ε, διακυβεύεται εδώ η δική μας αξιοπιστία. Το σύστημα ETS εκπομπών και πορείας ε, είναι πρωτοποριακό και το καλύτερο στον κόσμο, αλλά βεβαίως χρειάζεται και μεταρρύθμιση. Ελπίζω να συμφωνήσουμε για τη μεταρρύθμιση αυτή και να ε, είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε αυτή την υπόθεση υπό λετονική προεδρία, εφόσον έχουν γίνει πρόοδοι υπό την Ιταλική παρούσα προεδρία. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει ένα ξεκάθαρο τοπίο για όλους, ξέρει ο καθένας πώς θα κανονίσει την πορεία του. Η COP16 πλέον στην Κανκούν του Μεξικό ε, είχε αποφασίσει ε, και δεν έχουμε κάνει έκτοτε ε, σημαντική πρόοδο. Τελειώνει ο χρόνος και έχει έρθει ο χρόνος για δράση και για βήματα προς τα εμπρός. Ευχαριστώ πολύ. for... Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Συνάδελφος Τζο Λέν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορισμένοι εξημών ήταν ήδη στην Κοπενχάγη, στην ΚΟΠ. Και ζήσαμε τότε την απογοήτευση. Μετά δηλαδή από τις πολλές προσδοκίες τελικά δεν καταλήξαμε πουθενά. Αυτό δεν επιτρέπεται να μας ξανασυμβεί στο Παρίσι. Θεμέλιο για την επιτυχία είναι να είναι επιτυχής η έκβαση της διάσκεψης κορυφής της Λίμα να δοθούν μέσω αυτής τα στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν την παγκόσμια συμφωνία στο Παρίσι. Από το σχέδιό μας εσείς αναφέρατε μερικά θεμέλια, τα γνωρίζω καλά όλα. Χρειαζόμαστε παγκόσμια διαβεβαιώσεις από όλες τις χώρες δηλαδή για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Η διάσκεψη κορυφής της Νέας Υόρκης χθε ήταν χρήσιμη γιατί είδαμε τώρα ότι και οι μεγάλες χώρες εκπομπών όπως Κίνα και Ενωμένες Πολιτείε, είναι διατεθειμένες να κάνουν μια προσπάθεια, να καταθέσουν και αυτές τα χαρτιά τους δηλαδή. Ο, ρόλος, ο, ο λόγος για τον οποίο δεν καταλήξαμε σε αποτέλεσμα στην Κοπενχάγη ήταν διότι έπαιξε ένα πινκ-πονγκ Κίνα και Ενωμένε Πολιτείε. Οι Ενωμένε Πολιτείε είπαν αν η Κίνα δεν κινηθεί δεν κινούμεθα κι εμεί. Η Κίνα είπε οι Ενωμένε Πολιτείε είναι αυτέ που ρηπαίνουν περισσότερο και ούτω καθεξή. Αυτός ο γόρδιος δεσμός λύνεται τώρα. Όλες λοιπόν οι χώρες, σχεδόν, αν όχι όλες οι περισσότερες, πάνε να συμφωνήσουν, πάνε να συμμετάσχουν σε μια συμφωνία για την ανάγκη να διατηρηθεί η αναθέρμανση του κλίματος σε ποσό, σε λιγότερο των δύο βαθμών Κελσίου. Αν εξετάσει κανείς οριστικά, τις, ε, ιστορικά μάλλον τις επιβαρύνσεις, θα δει ότι οι βιομηχανικές χώρες έχουν επιβαρύνει πολύ περισσότερο και οι αναπτυσσόμενες χώρες αρχίζουν τώρα να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Θα κάνουμε λοιπόν αναγκαστικά περισσότερες προσπάθειες. Έτσι θα γίνει στη Λίμα, έτσι θα γίνει και στο Παρίσι. Και ερχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να έχουμε και να δείξουμε την θέληση να εγκρίνουμε του τρεις στόχους του κλίματος. Ο Κοινοβούλιο είπαμε τι θέλουμε. Τρεις δεσμευτικούς στόχους και όχι μονάχα ένα δεσμευτικό στόχο. Ελπίζω λοιπόν να τα καταφέρουμε. Το δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ψάξει να εξασφαλίσει τη μεγάλη εκείνη πλειοψηφία που θα επιτρέψει να πιέσει μετά την Κομισιόν και το Συμβούλιο προς την ίδια κατεύθυνση. Μένει και το ερώτημα της χρηματοδότησης. Αυτό είναι το περίφημο μαύρο κουτί. Ούτε στην Νέα Υόρκη είδα να λένε από που θα βρουν τα 100 δισεκατομμύρια. Αναμένουμε ακόμα τις καινοτόμες ιδέες διότι είναι αρκετά σφιγμένοι οι προπολογισμοί μα. δεν θα βρούμε λοιπόν εύκολα τα 100 δισεκατομμύρια, θα πρέπει να βρεθούν και από τον ιδιωτικό τομέα, κοινοπραξία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα δηλαδή, για να δούμε πώ θα χρηματοδοτήσουμε τα έργα που είναι απαραίτητα. Θα θυμίσω εδώ μονάχα τι επιδοτήσει για δραστηριότητε βλαπτικέ του κλίματο. Μέγα θέμα αυτό και στην Ευρώπη βεβαίω και στον κόσμο. Πρέπει να προχωρήσουμε και στο τοσί αυτό και να πάψουμε να χρηματοδοτούμε πράγματα που δεν θέλουμε πλέον. Μόλις ήρθα από μια εκδήλωση της Ισαβέλα Λεβίν για το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική, όπου άκουσα ότι ορισμένες τράπεζες όπως η Union Suisse αλλά και η Γερμανική Τράπεζα και άλλες είπαν ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν πλέον εργοστάσια παράγουν ενέργεια από άνθρακα. Το ίδιο πρέπει να εξετάσουν και οι χώρες πλέον να μειώσουν τις επενδύσεις σε τέτοια έργα και να χρηματοδοτήσουν άλλα τα οποία να είναι χρήσιμα. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε σωστή βάση, θα δούμε πώς θα προχωρήσει η συζήτηση και ποιες τροπολογίες τελικά θα υποβληθούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Ντάνκαν, για το ECR έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Το ECR καλωσορίζει το σχέδιο ψηφίσματος. Πιστεύουμε ότι βοηθάει να επιτευχθεί πρόοδος. Έχω κάποια σχόλια. Όσον αφορά τι ελπίζουμε να πετύχει το σχέδιο κειμένου τη συμφωνία. Πρώτα απ' όλα, αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα των χωρών, την εξέλιξή του και μελλοντικέ δυνατότητε. Και αυτό είναι το βασικό, ο πυρήνα πρέπει να έχουμε φιλόδοξες υποχρεώσεις και δίκες για όλες τις χώρες, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Και θα πρέπει να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο των δύο βαθμών. Μπορεί να είναι εφικτό, πρέπει να είναι εφικτό. Πρέπει να είναι αυστηροί κανόνε για να μπορούμε να βλέπουμε ποια πρόοδο έχει επιτευχθεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε ισχυρισμού χωρί να μπορούμε να του προσμετάμε ισχυρισμού. Πρέπει να υπάρχει περιοδική ακαιρεότητα και να γίνεται έλεγχο σε όλε τι χώρε, και στον ανεπτυγμένο και στον αναπτυσσόμενο. Και τέλο θα πρέπει να δώσουμε στηρίξη εκείνου που θα πρέπει να ε, μειώσουν τι εκπομπέ. Είναι σημαντικό για πολλέ χώρε, πολλά πρέπει να κάνουμε εδώ, να βοηθήσουμε τι πιο φτωχέ και τι πιο ευάλωτε ε, να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και στις απαιτήσει. Έχουμε πέντε στόχους που θα ήθελα να πετύχουμε ή να θέσουμε μάλλον από τη συζήτηση. Πρέπει να έχουμε συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο οι χώρε μπορούν να προωθήσουν τι δικέ του υποχρεώσει, να καταλάβουμε τι ακριβώ δεσμεύονται να κάνουν. Πρέπει να έχουμε συμφωνήσει όσον αφορά τα βασικά στοιχεία διαπραγματευτικού κειμένου. Θα είναι στο επίκεντρο τη προόδου αυτό. Πρέπει επίση, πιστεύω, όσο προχωρούμε προ το κείμενο του 2015 να εξετάσουμε κάποια σημαντικά θέματα περιστρέφονται γύρω από το καθεστώ, αλλαγή καθεστώτο, αλλαγή κλίματο, χρηματοδότηση που ενδείκνεται, ε, προκλήσεις για την αναγκαία προσαρμογή, τεχνολογία και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πραγματικότητα, όχι απλώς σε ένα εργαστήριο ή σε μια αίθουσα διδασκαλίας. Αν τα κάνουμε αυτά μπορούμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο και πρέπει να δούμε και τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι βασικό στοιχείο. Ζητάμε πάρα πολλά από τον κόσμο, πρέπει να είστε σίγουροι ότι θα μπορούμε να δεσμεύσουμε τα αναγκαία χρήματα για να πετύχουμε τους στόχους. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι τομείς όπου πιστεύουμε ότι το σχέδιο ψηφίσματος θα πρέπει να προσαρμοστεί θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία. Παράγραφος 1 βέβαια εδράζεται επί προηγουμένων ε, ψηφισμάτων ΚΟΠ, αλλά θα ήταν καλό να δείτε την ακμή, το ανώτατο σημείο του 2015. Δεν είναι κάτι εφικτό. Ακόμα ζητάμε και για μια μέγιστη τιμή το 2020 και αυτό είναι πολύ φιλόδοξο και αυτό το σημείο μπορεί να σε οδηγήσει σε δύο βαθμούς. Καλύτερα στο 50% μείωση μέχρι το 2050 να συγκεντρωθούμε. Ε, αυτή θα κάνει τη διαφορά. Πρέπει να διευκρινίσω στην παράγραφο 2 ότι αναμόρφωστε σε ε, μειώσεις και όλες οι μεγάλες οικονομίες θα πρέπει να εφαρμόσουν τα δικά τους ε, σχέδια για τη μείωση, να γίνει μείωση πιο πριν. Παράγραφος 5 θα πρέπει να λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες για συμμόρφωση και όχι για ένα καθεστώς για συμμόρφωση. Αυτό θα βοηθά στην, ε, στο διάλογο. Πρέπει να δούμε και νέα διατύπωση θα τονίζει την προσαρμογή που θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της νέας συμφωνίας, η προσαρμογή. Με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις πιστεύω ότι σημειώνουμε σημαντική πρόοδο στην αίθουσα αυτή προς σημαντική συμβολή στις γενικές συζητήσεις που θα διεξαχθούν στη Λίμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ σίγουρα. Θα λάβουμε διάφορες τροπολογίες από το ECR υπό το φως των παρατηρήσεων που ακούσαμε. Για τους φιλελεύθερους. Συνάδελφε Γκερμπραντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε στον αθλητισμό. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι χειροπιαστό, που είναι η φυσική κατάσταση, η φόρμα. Δεν είναι μόνο φυσική, μπορεί να είναι και πνευματική κατάσταση, είναι μια γενική κατάσταση. Καμιά φορά έχει την αίσθηση ότι είναι σε πλήρη φόρμα ο αθλητής ή η αθλήτρια και έχει πολύ κακές επιδόσεις. Στην πολιτική ε, αυτό ε, μεταφερόμενο ονομάζεται συγκυρία, momentum. Το 2009 στην Κοπενχάγη θεωρήσαμε ότι εκείνη ήταν η ώρα πραγματικά για να έρθει μια διεθνή συμφωνία στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Τεράστια απογοήτευση όμως ακολούθησε. Ορισμένοι από εμάς ήμασταν εκεί παρόντες και κάποιοι άλλοι μπορεί να το παρακολούθησαν απαλού. Έκτοτε δεν έχει ξαναδημιουργηθεί αυτή η ευκαιρία ε, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτή τη φορά στο δρόμο για το Παρίσι και περίεργος ο πιο ε, κοντινός δρόμος από εδώ στο Παρίσι είναι μέσω Λίμας, περίεργο πράγμα, και έχω σιγά σιγά την αίσθηση ότι ξανάρχεται αυτή η ευκαιρία, για διάφορους λόγους. Ο είναι αρνητικός. αισθανόμαστε ότι επήγει όλο και περισσότερο η κατάσταση και κινδυνεύει να μας ξεφύγει. Αυτά γίνονται ερήμην ημών. Πριν από δύο εβδομάδες ε, ο Οργανισμός Μετρολογίας στην Γενέβη ε, εξέδωσε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι υψηλότερε από ποτέ. Είδαμε κάποιες αναφορές και εκθέσεις από τη ΣΥΠΑ και αλλού ε, για θεομηνίες οι οποίες άμεσα πλέον συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Αυτός είναι ένας από, το, από τους λόγους που μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι είναι όλο και πιο επίγουσα κατάσταση. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι αρχίζει να κινείται λίγο περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας, πολύ περισσότερο από ό,τι στην Κομπεχάγη. Ε, οι εταιρείε επενδύουν όλο και πιο πολύ στην καθαρή τεχνολογία. Μια ε, χώρα όπως η Κίνα βλέπει μια τεράστια αγορά καθαρής τεχνολογίας να αυξάνεται και απομακρυνόμαστε από επενδύουν ε, στα ορυκτά καύσιμα. Κάποια Αμερικανικά ε, ε, πανεπιστήμια και συμφέροντα φεύγουν. 50 δισεκατομμύρια ε, δολάρια βγάζει σε επενδύσεις η οικογένεια Ροκφέλερ από τους υδρογονάνθρακες και τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, βλέπουμε έκθεση με την έκθεση να δείχνει ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η επιλογή μιας οικονομίας που παράγει λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα δεν είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ε, ε, ε, βιομηχανίας. Το αντίθετο θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα. Λοιπόν, βλέπω να ξανάρχεται τώρα η ευκαιρία αυτή. Η σύνοδο κορυφής του Ban ήταν εθαρρυντική. Έχω ακούσει εθαρρυντικά όχι μόνο από διάσημους Αμερικανούς ε, ηθοποιούς, αλλά και από αγνώστους ε, ή και από σήμους ή ακόμα και από τον πρόεδρο Ομπάμα και άλλους. Βλέπουμε η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να συναντώνται για να αντιμετωπίσουν από κοινού την κλιματική αλλαγή και θα πρέπει να προσέξουμε πραγματικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μείνουμε πίσω για να μην υπολοιπόμεθα αυτών των προσπαθειών. Ελπίζω ειλικρινά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 24 Οκτωβρίου να μην υποκριθεί ε, ε, ότι απλώς αποφασίζουμε και δεν κάνουμε τίποτα. Η Λίμα είναι ένα βήμα πριν το Παρίσι, Πρόεδρε, και ελπίζω να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ε, επιρροή μας για να επηρεάσουμε θετικά τις εξελίξεις και του χρόνου να πάρουμε τις δέουσε αποφάσεις στο Παρίσι. Ευχαριστώ. E Ευχαριστώ. Η κυρία Ροντρίκες Κουρμπιό έχει το λόγο για την ΚΟΕ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εσείς ε, γνωρίζετε μεταξύ σας εδώ και καιρό. Έχετε συζητήσει ε, για προηγούμενες συνόδους κορυφής. Εγώ την πρώτη φορά ε, που βρίσκομαι σε ένα δημόσιο θεσμικό όργανο είμαι εδώ, αλλά έχω ζήσει από τα κοινωνικά κινήματα της Συνόδου Κορυφής. Με σύνοδο τη Σύνοδο προσπαθούσαν να φέρουν τις προτάσεις τους εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Σήμερα το πρωί Είμαι καινούρια βέβαια, αλλά μαθαίνω πολύ και γρήγορα και ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συζήτηση ε, για την ε, εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Και βλέπω πολλά νεύρα, λόμπι, ε, email. Ορισμένοι τα βλέπουν αυτά με κάποιο φόβο, άλλοι με κάποια συντροφικότητα. Ο φόβος πάντα επιβάλλεται ως εκβιασμός για την ε, υγεία και για την απασχόληση. 400.000 ε, ε, το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη σε μια διαδήλωση διαμαρτυρήθηκαν για την κλιματική αλλαγή και προσπάθησαν να φέρουν στη Σύνοδο Κορυφής που συγκάλεσε ο Μπάνκι Μούν ένα μήνυμα και τους ανήθηκαν την είσοδο. 19 ε, συσκέψεις και διασκέψεις του ΟΗΕ έχουν γίνει, ε, ντουζίνες ολόκληρες προπαρασκευαστικές, τα περισσότερα κράτη-μέλη ε, και της Ένωσης δεν ποτάρουν απλώς την αδράνεια, αλλά υπερασπίζονται τη βιομηχανία. Λες όλα αυτά να ήταν πάντα αρμονικά με τα δικαιώματα και τη ζωή των ανθρώπων. Πολύ ωραία λόγια έχει το ψήφισμα βρήθη και δεσμεύσεις. Είδαμε όμως ότι ψηφίσαμε πριν από λίγο για ε, το να είναι δωρεάν οι εκπομπές στον ΥΠΟ Το Δεκέμβριο θα συστηθεί η Σύνοδος των Λαών που θα εκπροσωπούνται οι λαοί που πλήττονται και οι κοινότητες ε, από την κλιματική αλλαγή παράλληλα με τη σύνοδο του ΟΗΕ και ζητούν μια συμμετοχική, δημοκρατική και δεσμευτική συμφωνία με βάση τις κοινέ ευθύνε, την ισότητα, κοινέ μένα διαφοροποιημένες και κάτω από 1,5 ε, βαθμό θέλουν, όχι 2 βαθμούς, να ξεφύγουμε από τα ε, ορυκτά καύσιμα, το πετρέλαιο, την υδρορογμάτωση, να προχωρήσουμε στις ανανεώσιμες, στην τοπική παραγωγή και κατανάλωση, τοπική παραγωγή παντού για να ε, καλύπτονται οι τοπικές διατροφικές ανάγκες. Αυτό το πράγμα λέγεται διατροφική κυριαρχία. αν δίνουμε τζάμπα το δικαίωμα στις εταιρείες να συνεχίσουν να ρηπαίνουν ή να αυξάνουν το τιμολόγιο ε, του ηλεκτρικού, ενώ δεν τους κοστίζει τίποτα, την πληρώνει ο καταναλωτής, δεν πάμε καλά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτά που πρότεινε δεν έχει βάση ούτε επιστημονικά και αν δεν μπορεί να αντισταθεί. Ε, τι η Κομισιόν είναι αυτή που δεν μπορεί να αντισταθεί στι εταιρείε και στα συμφέροντά του. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τους πρασίνους ε, συνάδελφε ότι είχε το λόγο. Ευχαριστώ και με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούω από τους συναδέλφους μου πόσο πολλοί επιθυμούν να φτάσουμε σε μια παγκόσμια συμφωνία. Βέβαια, ακούω όλες αυτές τις ώρες τις ιστορίες και αισθάνομαι τον πειρασμό να γίνω κοινικός. Τέλος πάντων, ακούω τις ε, ε, υποσχέσεις και τις πιστεύω. Ας αγωνιστούμε υπέρ μιας παγκόσμιας συμφωνίας. Πραγματικά όμως να αγωνιστούμε, γιατί είναι ενδιαφέρον να διαπιστώσει κανείς ότι το 2009 ήταν η Κοπενχάγη και θυμούμε καλά που είχαμε τις κέρυες εκείνες συζητήσεις στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, εκεί το 2009 περίπου, πόσα χρόνια έχουν περάσει, είχαμε όλους τους πρωθυπουργού που πήγαιναν στην Κοπενχάγη και μας έλεγαν ότι είναι στο top της ατζέντα τους και χρειάζεται να αναλυφθεί δράση. Όλοι οι πολιτικοί τέτοια λόγια χρησιμοποιούσαν. Και μετά από αυτό ήρθε η αποτυχία και τους έλειψε και η πρόθεση. Από τότε δεν μιλήσαμε πολύ για το κλίμα και σίγουρα δεν μιλήσαμε στις κέρυες στιγμές ή στις ε, ώρες εχμής της Ολομέλειας. Μιλούσαμε καμιά φορά τη Δευτέρα το βράδυ, σαν δήθεν να μην αλλάζει πλέον το κλίμα. Από τη μια μεριά δηλαδή έχουμε τους πρωθυπουργούς που λένε ότι είναι μεγαλύτερη πρόκληση και τέσσερα χρόνια μετά κάνουν σαν να μην υπάρχει αυτή η αλλαγή του κλίματος. Και σαν να μην υπάρχουν και οι να μην, ε, αυξάνονται και οι ανανεώσιμες. Η κατανάλωση ανανεωσίμων κάθε χρόνο στην Ευρώπη αυξάνεται κατά 5%. Αν δει κανεί αυτέ τι εξελίξει, είναι πραγματικά πολύ παράξενο που τώρα, μια πενταετία μετά την Κοπενχάγη, συζητούμε και πάλι και λέμε Αχ, τι είναι καλό νέο που σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει μια όθηση το πράγμα. Καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι η πολιτική και εννοώ και εμάς που είμαστε εδώ, αν πραγματικά εννοούμε αυτά που λέμε στα σοβαρά. Και πιθανώς, αν τα ελοποιήσουμε αυτά, να αυξήσουμε λίγο και την εμπιστοσύνη του κόσμου στους πολιτικούς. Διότι διορωτώμεθα γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν πλέον στους πολιτικούς, ίσως πρέπει να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε και τη συνέπειά μας. Δεν θα μείνουμε λοιπόν με σταυρωμένα τα χέρια, θα αγωνιστούμε, να περάσουμε και από το Παρίσι, να πάμε στο Περού. Έγιναν εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο και στο Άμστερνταμ έκανα και εγώ πορεία και είχα την εντύπωση ότι ο κόσμος θέλει πραγματικά την αλλαγή και ζητεί το κοινό από την πολιτική ελίτ πραγματικά να αρχίσει να δρά και να υλοποιεί τις υποσχέσεις της. Πρέπει να τα αποκριθούμε λοιπόν οι πολιτικοί, διότι αλλιώς όλοι οι λόγοι αυτοί δεν έχουν μεγάλη αξία. Το μεγάλο ερώτημα για την Δήμα είναι βέβαια η αξιοπιστία της Ευρώπης. Και θέλω να ρωτήσω εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που φτιάχνει ωραία φυλάδια και τα τυπώνει για να δείξει τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι καταπληκτικά πράγματα που κάνει όντας πρωτοπόρα στον κόσμο. Αλλά ας διαρωτηθούμε Ας πάμε σε μια αναπτυσσόμενη χώρα που ακούει τον Μπαρόσο να λέει στη Νέα Υόρκη ότι θα φτάσουμε στο μείον 80%, στο μείον 90% μέχρι το 2030. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση για μείον 95%. Να αφήσετε λοιπόν τις ανοησίες αυτές, βγάλτε από το λόγο του Μπαρόσο τις ανοησίες αυτές. Ας πει μείον 80 και μετά να δούμε ίσως αν μπορεί να υπάρξει κάποια αξιοπιστία. Αυτό όμως ισχύει και για μας, γιατί τα πιο, πολλά, πιο σημαντικά πράγματα είναι η αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας των εκπομπών. Σήμερα υπάρχει μια πλειοψηφία, διαμορφώνει μια πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να φτάσει η τιμή του τόνου του διοξιδίου του άνθρακα στα 30 δολάρια. Να αγωνιστούμε όμως για να γίνει αυτό. Όχι πάλι καινούριε φραστικές φιωριτούρες που δεν ενοχλούν καθόλου την βιομηχανία. Και τέλος το μέγα θέμα είναι η χρηματοδότηση. Εδώ και μια δεκαετία υποσχόμεθα ότι μέχρι το 2020 θα διαθέσουμε 100 δισεκατομμύρια δολάρια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κάθε χρόνο όμως, κάθε χρόνο όμως αποφεύγουμε να το πράξουμε. Πώς λοιπόν να πιστέψουν οι αναπτυσσόμενες χώρες ή ότι οι αναπτυγμένες χώρες θα τους δώσουν όντως τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2020. Αν δεν τροπάξουν αυτό, τότε οι αναπτυσσόμενες χώρες καλά θα κάνουν να πούν ότι δεν τους πιστεύουμε τους Ευρωπαίους. Λόγια λένε και δεν κάνουν τίποτα. Και το Παρίσι θα είναι άλλη μια Κοπενχάγη, άλλη μια αποτυχία. Έχουμε 15 μήνες, ας το παλέψουμε, ας αγωνιστούμε, Αλλιώς θα σταματήσουμε να εκφωνούμε τέτοιους λόγους. Ευχαριστώ. Η FTD Ματζουρόνη, συνάδελφε Ματζουρόνη, για το λόγο. Thank you, Chairman. Αγαπητοί συνάδελφοι, στη Λίμα, την πρωτεύουσα του Περού, θα διεξαχθεί αυτή η διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή είναι 20. Καταρχήν, είναι ο τελευταίος σταθμός αυτός πριν την κρίσιμη συνεδρίαση στο Παρίσι το 2015. Η διάσκεψη θα πρέπει να σκιαγραφίσει τα βασικά χαρακτηριστικά της Παγκόσμιας Συμφωνίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η διάσκεψη επίσης θα πρέπει να καταλήξει σε κάποιο σχέδιο κειμένου για τη συμφωνία. Συνάδελφοι, ελπίζω να θυμόσαστε τι έγινε στην 19η διάσκεψη στη Βαρσοβία. Συμμετείχα εκεί σαν εκπρόσωπος της Λιθουανίας που είχε τότε την ε, Προεδρία. Αν δούμε ποια ήταν, ποιες ήταν οι ελπίδες και ποια ήταν τα αποτελέσματα, είναι σαφές ότι ε, τα αποτελέσματα στη Λίμα δεν θα είναι καθόλου εύκολα να τα πετύχουμε. Οι χώρες στη διάσκεψη θα πρέπει να έρθουν με συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και οι υποχρεώσεις που έχουν αναλυφθεί θα πρέπει να είναι πρόδρομοι των υποχρεώσεων που θα αναλυθούν το 2015 στην 21η ΚΟΠ. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι από μόνη της η ευρωπαϊκή προσπάθεια δεν αρκεί. Ποιο είναι ο κίνδυνος? Ότι μετά το 2020 ίσως να ξεπεράσουμε τα ασφαλή όρια για την αλλαγή του κλίματος. Γι' αυτό κάθε χώρα πρέπει να κάνει τη δουλειά της να τακτοποιήσει τα του οίκου της. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα σχέδια δράσεως με συγκεκριμένες υποχρεώσεις από κάθε χώρα, ούτω ώστε να καλυφθούν τα διάφορα κενά και οι διαφορές που υπάρχουν. Χρειάζεται ένα παγκόσμιο σχέδιο, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα αφορά όλες τις χώρες του κόσμου. Όλες οι χώρες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι πρέπει να καλυφθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ επιστημονικής έρευνας από τη μια και πραγματικής κατάστασης από την άλλη. Οι δεσμεύσεις να μειωθούν τα αέρια του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 και ποιες είναι οι πραγματικές εκπομπές, υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο υποσχέσεων και πράξεων. Και οι τάσεις που έχουμε τώρα δεν αρκούν για να πετύχουμε το στόχο των δύο βαθμών πρέπει να σπρώξουμε τις άλλες χώρες, οι ιδιωτικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικοί φορείς, όσοι ενδιαφέρονται να βρεθεί κοινό τόπος, ούτω ώστε να συνεργαστούμε, γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σουίκα, συνάδελφε Σουίκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω κι εγώ σε αυτή τη συζήτηση γιατί χαίρομαι πάρα πολύ που στη δική μας Επιτροπή είναι ένα θέμα που κυριαρχεί η κλιματική αλλαγή. Τώρα προτείνουμε ένα νέο ψήφισμα αρκετά φιλόδοξο. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να μειωθούν κατά 50% οι εκπομπές ε, των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020. Και λέμε ότι τότε θα φτάσουμε στο επίπεδο το 1990. Έχουμε δεσμευτεί να μειώσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, τηρήσουμε τα όσα έχουμε υποσχεθεί μέχρι το 2020 και σε σχέση με τη συμφωνία της Κοπεχάγης. Πρέπει να σας πω ότι μου παρούσα, προσωπούσα τότε το Συμβούλιο της Ευρώπης και κάποιες περιφερειακές αρχές και είναι πολύ απογοητευτικό το γεγονός ότι ήταν μια τρύπα στο νερό αυτή η συμφωνία ελπίζω και εύχομαι να γίνουν πολλά περισσότερα στο Παρίσι. Καλώς ορίζω και τη χθεσινή εκδήλωση και σύνοδο κορυφή στη Νέα Υόρκη. Προσβλέπω στη Λίμα το Παρίσι και ελπίζω το 15 το Παρίσι να καταφέρει να πετύχει όλους τους στόχους που συζητούμε. Για να μην μιλάμε μόνο πολύ χωρίς να εφαρμόζουμε τίποτα. Σε εμάς εναπόκειται και στα κράτη-μέλη να συνεχίσουν όλες αυτές τις δραστηριότητε να γίνουν οικονομικές συνεισφορές από πλευράς των κρατών μελών και είμαι επίσης και υπέρ ισχυρής παρακολούθησης, ε, αναφοράς και ε, επαλήθευσης για να υπάρχουν έλεγχοι και επαληθεύσεις. Και επίσης να αναφερθώ και στι τιμές του διοξιδίου του άνθρακα το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ορισμένοι έχουν πολύ στεναρές απόψεις, άλλοι λιγότερο ε, δυνατά ε, το φωνάζουν. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Μιλούμε για μεγάλες παγκόσμιες ε, χώρες, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει και με αυτούς να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε, αλλά να μην λησμονούμε και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πολύ συχνά τις κατηγορούμε και τελικά τις τιμωρούμε κιόλα. γιατί ε, δεν υπάρχουν οι πόροι. Εγώ είμαι από την Κροατία. Έχουμε υποστεί τρεις μεγάλες πλημμύρες πρόσφατα. Δεν έχουμε τα χρήματα για την ανοικοδόμηση της χώρας και την αντιμετώπιση των ζημίων. Επίσης μιλήσαμε για την αεροπορία, για την αυσιπλοεία. Θα πρέπει ε, όλα αυτά να εφαρμοστούν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Πίτερ έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσοι εργάστηκαν και πολύ σκληρά στην εκπόνηση του σχεδίου ψηφίσματος. Σήμερα το μεσημέρι αναφέρθηκε σε αυτό ο Γιολάινεν σε μια εκδήλωση που ε, διοργάνωσε μια συνάδελφος και κάποια άλλη βουλευτές θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Δεν είναι αδιάφορο το πότε θα αρχίσουμε να προστατεύουμε το κλίμα και με ποια ταχύτητα. Δεν είναι τυχαίο. Στα οικοσύστημα υπάρχουν κάποια καμπανάκια που χτυπάνε όταν δεν ε, αρχίσεις να μειώνεις τις εκπομπές εγκαίρως. Κάποια στιγμή ε, γίνεται μια καταστροφή που είναι ανεπανόρθωτη. Παράδειγμα, απλό. Στη μεταβατική ζώνη προς την Αρκτική, τη Βόρεια Ευρώπη κυρίως, αλλά και στη Ρωσία, υπάρχουν τεράστιες ποσότητες ε, ε, μεθανίου, ε, αερίου, που είναι κλεισμένες, εγκλωβισμένες μέσα στους αιώνιους πάγους. Ε, και αν λιώσουν ε, οι πάγοι ελευθερώνεται τέτοιο μεθάνιο ε, και που θα είναι άνευ η διαδικασία αυτή και δεν πάνε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να εξοικονομούν όσο διοξίδιο του άνθρακα θέλετε. Για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Γιατί κάποια στιγμή είναι πολύ αργά και το ρολόι, το, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ε, ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε 100 χρόνια να έρθει η τεχνολογία που χρειαζόμαστε για να τα διορθώσουμε. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, 7-8, αυτές οι λεγόμενες ορολογιακές βόμβες στα οικοσυστήματα, tipping points, ε, που κινδυνεύουν να εκραγούν και το θέμα είναι πραγματικά πάρα πολύ επίγον. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε μία διεθνή συμφωνία η οποία σίγουρα δεν θα είναι τέλεια. Αν μπορούσε ο καθένας από εμά χωριστά να συντάξει και αυτή τη συμφωνία, ε, θα ήταν πολύ πιο εύκολο από το να καταφέρεις να φέρεις σε μια συμφωνία όλες τις χώρες του κόσμου. Να μην έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις, παρόλο που η επιστήμη τα λέει αυτά και φωνάζει αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί είναι πολύ μεγάλες και πολλές οι διαδικασίες που χρειάζονται και πιστεύω ότι θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Είναι πολύ σημαντικό και σήμερα το πρωί το είπα. Το άφησα να εννοηθεί για το ρόλο της βιομηχανίας και χαίρομαι που κερδίσαμε την ψηφοφορία για το carbon leakage, ε, αλλά θέλω να απευθύνω μια έκκληση στη βιομηχανία. Δεν επιτρέπεται να λέει η βιομηχανία, κάντε εσείς ε, η πολιτική παγκόσμια συμφωνία και αυτή είναι παγκόσμιες εταιρείε. Η χημική βιομηχανία ε, στην Ευρώπη έχει εργοστάσια και στις Ηνωμένες Και έρχονται και λένε, κάνει προτάσεις ο Ομπάμα και τις υποστηρίζουμε. Μα το θέμα είναι να υπάρχει παγκόσμια συμφωνία που να λύνει όλα τα προβλήματα και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Λέω όμως με κάθε προσοχή προς τις ΜΚΟ και στους πράσινους φίλους μας ο βασικός ρόλος των ΜΚΟ και των Πρασίνων δεν είναι να κάνει όλο και περισσότερα η Ευρώπη και να το λέμε δέκα φορές συνέχεια. Χρειαζόμαστε παγκόσμιες λύσεις. Δεν αρκεί η Ευρώπη. Γι' αυτό καλωσορίζω πάρα πολύ τη δέσμευση των ΜΚΟ, τις ξέρω πάρα πολύ καλά, ας πούμε την κοινωνία των πολιτών ε, στην Κίνα. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και στην Κίνα ε, ότι υπάρχει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής Βεβαίως η Ευρώπη πρέπει να κάνει πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε από μόνοι μας τα πάντα. Μπορούμε να είμαστε ένα τμήμα της λύσης αν φανούμε έξυπνοι. Η κοινωνία των πολιτών είμαστε όλοι μας. Και θα πρέπει τώρα να ε, αδράξει την ευκαιρία να πιάσει το μπαλάκι που της πέταξε η διαδήλωση στη Νέα Υόρκη και οι πολιτικοί και καλλιτέχνες και άλλοι δημόσια πρόσωπα ε, ζητούν να αγωνιστούν ακόμα περισσότερο οι πολίτες προς αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει όλοι από κοινού να συνεισφέρουμε. Τελευταίο, ε, αεροπορία και ναυσιπλοεία, τα είπε και ο πρόεδρος, να πω λίγα πιο συγκεκριμένα πράγματα κι εγώ. Πιστεύω ότι οι αρμόδιοι υπεύθυνοι για την κλιματική αλλαγή που θα συναντηθούν στη Λίμα θα πρέπει να στείλουν ένα σαφές μήνυμα στον ΙΚΑΟ ε, και στον IMO, στο Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοής. Από το Κιώτο το 1997 και οι δύο οργανισμοί έχουν το καθήκον να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Εκεί να δείτε πόσο το συζητάνε. Αλλά έχουμε και το πρόβλημα ότι Έχουμε πάρα πολλά φρένα και χειρόφρενα, πολύ περισσότερα από ό,τι στον ΟΗΕ. Στον ΙΚΑΟ και το IMO φρενάρουν πολύ περισσότερο από ό,τι στη Λίμα και στο Παρίσι. Θα πρέπει λοιπόν και από τη Λίμα και από το Παρίσι να ζητήσουμε να πούμε ότι αν δεν λυθεί το πρόβλημα θα το λύσουμε αλλού αν δεν μπορείτε να λάβετε τις ευθύνες που έχετε υπομειστεί κύριε ΚΑΟ και ΆΕΜΟ το αναλαμβάνουμε εμείς και θα βρούμε τη λύση. Δεν χρειάζονται κλήσεις και τα λοιπά. Με προθεσμία, λοιπόν. Είτε θα το λύσετε, είτε θα το αναλάβουμε εμείς. Που σας το έχουμε αναθέσει και το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πίτερ. Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, λέει και Σπαρνιού, όπως ανέφθηκε, υπάρχει διαδοχή συνόδων κορυφής ε, για την αλλαγή του κλίματος, για την απειλή αυτή που βαρύνει τον πλανήτη. Όλοι φρονούν ότι είναι απογοητευτικό λυπηρό να μην μπορούμε να προχωρήσουμε καλύτερα, πιο μπροστά ήμουνα με τον πρόεδρο τον Τζο Λάινεν και πήγα στην Κοπενχάγη με μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής αυτής του περιβάλλοντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τέλος 2009 δεν έζησα μόνο μία απογοήτευση αλλά ε, παρέκκληση, αλλαγή πορείας όλων εκείνων που κήρυταν την ε, νίκη που διέβλεπαν μια συμφωνία επερχόμενη και τελικά επαναχωρήσαμε. Και όλες οι διεθνείς σύνοδοι κορυφής που γνωρίσαμε μετά το τέλος 2009 κάθε φορά ήταν μια απογοήτευση αυξανόμενη απογοήτευση έβγαινε από αυτέ. Όμω η Σύνοδο Κορυφή τη Νέα Υόρκη που προετοιμάζει τη Λίμα και το Παρίσι, προετοίμασε τη Λίμα και το Παρίσι, δεν παρέκλεινε από τον κανόνα, αλλά ταυτόχρονα ετέθη ένα κάπως διαφορετικό πλαίσιο. Και τολμώ να πω, αλλάζει το κλίμα. Είδαμε κινητοποίησει των πολιτών, αρκετέ δεκάδε πόλεων στον κόσμο κινητοποιήθηκαν. Είδαμε το Σαββατοκύριακο πάνω από 400.000 άνθρωποι στη Νέα Υόρκη κινητοποιήθηκαν. Απροσδόκητο να βλέπουμε τόσο κόσμο. Και κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε και μια κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση του οικονομικού κόσμου που φαίνεται να είναι έτοιμος να δράσει. Κάποια παραδείγματα. Ο Νίκολα ο οικονομολόγος, λέει ότι η καταπολέμηση της θέρμανσης, της θερμοκρασίας χάρη στον επαναπροσανατολισμό των επενδύσεων προς μη ανθρακοβόρες ε, τεχνολογίες ε, μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη χωρίς βλάβη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει ταυτόσιμη διαπίστωση. Λέει ότι αυτή η καταπολέμηση όχι μόνο δεν εμποδίζει την ανάπτυξη την οικονομική, αλλά αντίθετα τονώνει τη δημιουργικότητα και συνεπώς τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Στη Νέα Υόρκη ακούσαμε έναν ασιατικό ε, γίγαντα της οικονομίας, ε, χαρτοβιομηχανίας, ε, που προσπαθεί να, να κόβει λιγότερα δέντρα. Και άλλοι είπαν ότι θα σταματήσουν επενδύσεις όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα. Είναι έτοιμη η κοινωνία, ε, το είδαμε σε, στις διαδηλώσεις παντού στον κόσμο. Το περασμένο Σαββατοκυριακό ο οικονομικός κόσμος όλο και περισσότερο φαίνεται επίσης να ευαισθητοποιείται. Η τεχνολογία ε, ακολουθεί σε κάποιο ρυθμό. Ε, έχουμε τα φωτοβολταϊκά, αποθήκευση της ενέργειας, ευφυή δίκτυα, οπότε δεν μένει παρά μια πολιτική συμφωνία διεθνής, φιλόδοξη, που θα μπορεί να καθορίσει νέους κανόνες του παιχνιδιού όσον αφορά την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, ούτω ώστε οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις να γίνουν πιο αποδοτικές για το κοινό καλύτερες από τις επενδύσεις που έχουν στόχο άμεσο όφελος. Ιδού λοιπόν ο ρόλος που έχουμε σαν πολιτική να παίξουμε ε, όσον αφορά την ευαισθητοποίηση. Άκουσα κάποια λόγια σήμερα το πρωί στη συζήτηση που διεξήχθη όσον αφορά τις διαρροές του άνθρακα. Λοιπόν, ε, όπως και υπάρχουν λόγια, αλλά τίποτα δεν είναι δυνατόν σαν ε, χωρίς τις αποδείξεις. Ευχαριστώ και για αυτή την τελική, το τελικό που είπατε, που είναι κάτι σαν την αγάπη, πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Συνάδελφε Πάξο, για τους μη γεγραμμένους, ευχαριστώ. Το 2009 ήμουνα μέλος του Ευρωκοινοβουλίου για 10 μήνες και ήμουνα αναπληρωματικό μέλος της ΕΝΒΗ και ετοιμαζόμασταν τότε για τη Σύνοδο Κορυφή τη Κοπενχάγης. Πέντε χρόνια μετά έχω την εντύπωση ότι σταμάτησε ο χρόνο, σταμάτησαν τα ρολόγια. Ακούω τα ίδια πράγματα ξανά. Μου λέγουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα υπομισθούν κάποιε ευθύνε, θα καθορίσουν κάποιου φιλόδοξου στόχου. Αυτό είναι καλό, πάρα πολύ καλό. α δώσουμε το παράδειγμα. Αλλά ακούω του πράσινου και οι πράσινοι μιλάνε για πιο φιλόδοξου στόχου και η πλειοψηφία φαίνεται να τους υποστηρίζει. Και το ίδιο ακούγαμε και πριν την Κοπενχάγη. Ποιος είναι ο κοινό παρονομαστής, λαμβάνοντας υπόψη το ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα αρνούνται να συμμε... αρνήθηκαν να συμμετάσχουν την προηγούμενη φορά στη Νέα Υόρκη. Είχαμε τον Αλ Γκόρ που έκανε συζητήσεις, έγιναν συζητήσεις μεταξύ ΙΠΑ και Κίνας ποιος κερδίζει το χρυσό όσον αφορά τη ρήπανση, ποιος μολύνει περισσότερο, θα πρέπει να πάρουν και δύο ταργυρό γιατί και οι δύο είναι εξίσου κακοί. Ε, νομίζω ότι πραγματικό στόχο είναι να εξασφαλίσουμε ότι εκείνε οι χώρε θα υπομισθούν τι δικέ του ευθύνε. Γιατί στο κάτω-κάτω πρόκειται περί παγκοσμίου προβλήματο. Δεν έχει νόημα η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκουπίζει μπροστά στην πόρτα τη, να σκουπίζει την αυλή τη. Μιλάμε για ένα θέμα παγκοσμίου εμβέλεια. Εδώ μιλάμε για τι εκπομπέ και είμαστε υπεύθυνοι για 13% των εκπομπών αυτών. Αυτό είναι το μετικό μα. Ναι, βέβαια, πρέπει να πετύχουμε του δικού μα στόχου, να κοινοτοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών. Ναι, συμφωνούμε, αλλά ανακαλύπτουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που 500 εκατομμύρια ανθρώπους, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν πολιτικό βάρος αυτοί να κάνουν κάτι. Έχουν την πίεση των λόμπι να κάνουν κάτι. Και τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό μας Κοινοβούλιο, τι γίνεται με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους χρειαζόμαστε όλους να συμμετάσχουν, όλοι θα πρέπει τελικά να λογοδοτήσουν και να τηρήσουν αυτά που λένε διαφορετικά. Φοβούμε ότι δεν θα πετύχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε, θέλουμε κάτι δεσμευτικό, κάτι που μπορεί να υποπτευθεί και να εφαρμοστεί και να μπορεί να υπάρχει λογοδοσία και να κρίνονται αυτοί που δεν κάνουν ό,τι θα έπρεπε. Και θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι μεγαλύτεροι ρήπαντε, διότι διαφορετικά δεν θα πετύχουν τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ευχαριστώ. Ο αντιπρόεδρο Ζαβόρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αξιότιμοι συνάδελφοι. Σήμερα το απόγευμα αναφερθήκαμε εκτενώς στη σημασία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής που είμαστε, τι απομένει να κάνουμε θα μπορούσαμε να μιλάμε για διάφορα πράγματα, να μιλήσουμε για μια πράσινη οικονομία, μια πράσινη κοινωνία, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την πραγματική μετάβαση, πώς θα ήταν υποφελής αυτή για την οικονομία μας, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το πώς οι κοινωνίες μπορούν να αναδιαθρωθούν ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε βιώσιμη ενεργική πολιτική, κάτι πιο δημοκρατικό για τις κοινωνίες μας. Αλλά στο τέλος θα ήθελα να αναφέρω ένα σημείο και να το προσέξουμε παρακαλώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στα σχόλια του κυρίου Λίζε ο κύριος Λίζε έχει απόλυτο δίκιο, έθεσε ένα ζήτημα, δηλαδή το σημείο αλλαγής ισορροπίας. Είναι το σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό το κομβικό σημείο. Υπάρχουν καταστάσεις στο παγκόσμιο περιβαλλοντικό σύστημα ένα σημείο κομβικό πέρα το οποίο δεν υπάρχει ε, επιστροφή. Δεν μπορεί να ελέγξεις πλέον την κατάσταση. Ε, ε, μετά ο συνάδελφός μου ο κ. Λίζε αναφέρθηκε σε αυτά τα σημεία τα, τα κομβικά που ίσως να είναι κάπου στον ορίζοντα, στο μέλλον. Δυστυχώς όμως εγώ έχω κακά μαντάτα αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά τα κομβικά σημεία δεν στο μακρινό μέλλον, είναι πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά πίσω από τη γωνία. Και ο κύριος ε, Λίζε αναφέρθηκε στο θέμα της απελευθερώσεως μεθανίου των αιωνίων πάγων ότι στη Σιβηρία υπάρχει πολύ μεθάνιο αποθηκευμένο στου αιώνιου πάγου που θα μπορούσε αν λιώσουν οι πάγοι να απελευθερωθεί. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν είναι κάτι που θα συμβεί στο μακρινό μέλλον. Ήδη, τώρα, φέτο, είχαμε κάποια επιστημονικά άρθρα σύμφωνα με τα οποία αυτό συμβαίνει τώρα. Μιλάμε για κομβικό σημείο άνευ επιστροφής, μετά το οποίο σημείο το θέμα του κλίματος δεν θα μπορεί να, αλλάξει, δεν θα μπορούμε να κερδίσουμε πλέον τη μάχη. Αυτό θα πρέπει να καλύψουμε σαν άμεσο πρόβλημα. Σε 30 χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, με άλλα λόγια, η επόμενη γενιά δεν θα μας ρωτούν πλέον ε, ποια, ποιες ελαστικές ιδέες είχατε τότε, Καταλήξατε σε συμβιβασμό λογικό τότε. Μιλήσατε για την Κίνα, μιλήσατε για τη ΣΥΠΑ, τις ευθύνες που είχαν, ε, τα τονίσατε αυτά. Δεν είναι ένα ερώτημα θα μας ρωτήσουν ή τις επόμενες γενιάς θα μας πούνε. Κάνατε ό,τι μπορούσατε τα πάντα, ώστε να μπορέσετε να εγγυηθείτε έναν τρόπο ζωής αξιοπρεπή και αποδεκτό και βιώσιμο για όλους. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της δεν μπορεί να πολεμήσει αυτή τη μάχη, δεν μπορεί να την κερδίσει τη μάχη. Το είδαμε κατά το παρελθόν και εξακολουθούμε να το βλέπουμε τώρα. Είμαστε η πιο δραστήρια περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός φορέας στο παγκόσμιο προσκήνιο. Είμαστε εμείς που κάνουμε την πιο σκληρή δουλειά και μπορούμε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί, μπορούμε να είμαστε μεσολαβητές, να εξασφαλίσουμε το ότι η διεθνή κοινότητα θα υπομειστεί τις ευθύνες της, παραδεχτεί. Όλοι τελικά να υπομιστούν το βάρος τους. Δεν θα πρέπει μας λείψει το θάρρος. Δεν θα πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς που δεν είναι φιλόδοξοι. Διότι αν δεν είμαστε αρκετά γενναίοι, κανένας άλλος δεν θα κάνει τη δουλειά για μας. Κανένας άλλος θα είναι εκείνος που θα πολεμήσει τη μάχη τόσο σκληρά όσο μπορούμε εμείς. Αυτή είναι η δουλειά μας σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι η δουλειά μας σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είμαστε γενναίοι και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η Επιτροπή, η Επιτροπή Περιβάλλοντο, έχει ακριβώ αυτό το καθήκον. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν. Αυτή είναι η κλίση μα, η αποστολή μα. Και πιστέψτε μα, τα παιδιά σα και τα εγγόνια σα θα σα ρωτήσουν. Κάνατε τη δουλειά σα όπω έπρεπε. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε Ζαβόρ. Συνάδελφε Γκαρντίνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακολουθώ το ζήτημα αυτό από όταν μπήκα το 2008 στο Κοινοβούλιο, δηλαδή από την μυθική τώρα πια διάσκεψη της Κοπενχάγης, όπου πολλοί από τους παρόντες ήταν παρόντες και ζήσαμε μαζί πιστεύω αυτό το συλλογικό τραύμα, ας το αποκαλέσουμε έτσι, μια διάσκεψη που είχε παρουσιαστεί σαν η διάσκεψη που θα έπρεπε επιτέλους να επιλύσει το πρόβλημα με μια συμμετοχή των μίντια στο, στην γεγονός που ανέβασαν πολύ ψηλά τις προσδοκίες και όμως αντίθετα στο τέλος είχαμε κατάρρευση με τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε όλοι. Πρέπει να πω ότι σαν νεόφοιτη τότε με θαυμασμό έβλεπα τις προσδοκίες που ήταν τόσο ψηλές, διότι πριν μήνες ήμουνα στη Ουάσιγκτον και συναντήθηκα με γερουσιαστές που ήταν δημοκράτες, διότι οι ρεπουμπλικάνοι απέφευγαν να συναντηθούν. Γιατί για αυτούς η αλλαγή του κλίματος, πρωτόκολλο του Κιώτο και λοιπά ε, ακούγανε τέτοια πράγματα και ξεφεύγαν, την κάνανε από την άλλη. Και όλοι αυτοί είπαν ότι στην Αμερική ποτέ δεν θα μπορούσαν να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία στις ΗΠΑ. Και απέκλειαν ο Ομπάμα να μπορούσε να υπογράψει τη συμφωνία ε, όταν δεν υπήρχε κανένας νόμος στο Αμερικανικό δίκαιο που να μπορούσε να υποστηρίξει μια ενδεχόμενη υπογραφή. Θα ήταν κάτι αντισυνταγματικό για αυτούς μια τέτοια υπογραφή και με θαυμασμό έβλεπα αυτή τη διαφορά μεταξύ πραγματικότητας, ποια ήταν η αλήθεια και αυτή που περιγραφόταν. Και ανησυχούσα αρκετά βλέποντας μια Ευρώπη που από μόνη της ε, έβγαζε ένα παραμύθι, διγόταν ένα παραμύθι. Μετά ήρθε η κρίση και η κρίση δημιούργησε νομίζω μεταξύ πολλών άλλων δραματικών αποτελεσμάτων και μια αντιμετώπιση πραγματικότητας. Η Ευρώπη έγινε πιο συγκεκριμένη έπαψε να πιστεύει ότι για να είναι ηγέτης έπρεπε να είναι χιλιόμετρο μπροστά από τους άλλους διότι άμα τα έχεις μόνος σου και είναι πολύ πίσω όλοι οι άλλοι είσαι μόνος μοναχικός δρομέας και όχι ηγέτης της κούρσας και τελικά τώρα είμαστε πιο κοντά στην επίδευση της συμφωνίας. Στο Κιώτο είδαμε πώς κατέρευσε. Αν δεν φτάσουμε σε μια παγκόσμια συμφωνία, δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε, αλλά τα αποτελέσματα θα είναι πραγματικά μικροπράγματα. Δεν θα μπορούσαν να πετύχουν τίποτα από τους στόχους μας. Πιστεύω όμως η Τιλίμα και το Παρίσι Επιτέλους θα είναι οι στιγμές εκείνες κατά τις οποίες μια παγκόσμια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί και μάλιστα επειδή ε, εντάξει λέμε ότι πρέπει να είμαστε γενναίοι και να προχωράμε κλπ αλλά λέω ότι εμείς να γίνουμε όπως γίναμε ε, άνθρωποι που ε, μπαίνουν σε διάλογο. Αν μπορούμε να μειώσουμε 10% των παγκοσμίων εκπομπών ε, είμαστε στην, στη μειοψηφία. Μπορεί Μπορεί μια μειοψηφία να έχει αναλαμπές, να είναι πεφωτισμένη το 10%, αλλά 90% πρέπει να πιστούν οι εταίροι μας. Δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε. Πιστεύω και ελπίζω αυτή να είναι η επικοδομητική μας προσέγγιση και να καταφέρουμε τελικά να πετύχουμε τη συμφωνία, την παγκόσμια συμφωνία, τη σφαιρική συμφωνία που όλοι είμαστε πεπισμένοι διότι χρειάζεται. Είναι ο μόνος τρόπος αυτός να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα διαφορετικά θα είναι κάτι ανέφικτο. Πιστεύω ότι ποτέ όπως σήμερα δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις οι καλές. Και ελπίζω η δουλειά μας να οδηγεί σε επιτυχία. Και επιτέλους να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία παγκοσμίου επίπεδου που επιθυμούμε. Ευχαριστώ, Ελιζαμπέτα. Συνάδελφε Λόβιν, έχετε το λόγο. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που ήρθαν στην εκδήλωση που διοργάνωσα σήμερα μαζί με τον Γιώ Λάινεν και τον Πέτερ Λίζε. Ήδη αναφέρθηκε επανειλημμένα στη συζήτηση αυτή η εκδήλωση και επ' ευκαιρία θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους για το τι διεμήθη εκεί Είχαμε τέσσερις επιστήμονες κορυφές ε, σε θέματα πολικής επιστήμης και ωκεανογραφίας και μας εξήγησαν ε, ποια είναι τα πιο πρόσφατα ευρήματα ε, σχετικά με την κλιματική αλλαγή και πώς επηρεάζει τους ωκεανούς. Το είπε και ο συνάδελφος Γιαβόρ για τα σημεία που δεν υπάρχει επιστροφή Ας πούμε, στην αύξηση της στάθμης των ωκεανών, δύο είναι επιστημονικές ομάδες που κατέληξαν σε πολύ αντίστοιχα αποτελέσματα και τώρα το Μάιο οι ανακοινώσεις τους ε, δημοσιεύτηκαν από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και ένα της Καλιφόρνιας που έλεγαν ότι λιώνουν οι πάγοι στην Ανταρκτική και αυτές οι έρευνες αλλά και ανεξάρτητες έχουν ε, μελετήσει ε, το λιώσιμο των ε, παγετώνων ε, και ότι μέχρι και τέσσερα μέτρα θα αυξηθεί λέει η στάθμη των ωκεανών και αυτό είναι μη αντιστρεπτό και μη αναστρέψιμο. Μπορεί να μην γίνει τον παρόντα αιώνα και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο πιο άνετα αλλά αν δούμε την ταχύτητα που θα πάρει αυτό μπορούμε να το επηρεάσουμε η πολιτική απόφαση μπορεί κάπως να συγκρατήσει ε, αυτή την ορμητική εξέλιξη και το ρυθμό. Πάντως ότι θα γίνει, θα γίνει. Δεν ε, τίθεται θέμα και θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Τέσσερα μέτρα θα ανεβεί η στάθμη των ωκεανών. Υπάρχουν και άλλοι παγετώνες που ενδεχομένω να λιώσουν αλλού. Αν λιώσει όλο το στρώμα που καλύπτει την αντακτική θα φτάσει μέχρι και τα 55 μέτρα η στάθμη των ωκεανών προς τα πάνω. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές. Επίσης η οξύνωση των ε, ωκεανών είναι πάρα πολύ αρνητικό. Δεν είναι πρόβλεψη αυτό ούτε ε, τίποτα μαντικές. Ε, μέτρα με το pH στους ωκεανούς το οποίο μειώνεται. Ίσον όξινο και αν ε, ακόμα και με το στόχο του, των δύο βαθμών Κελσίου είναι πολύ ενισχυτικέ αυτές οι εξελίξεις όταν αφορά όλα τα θαλάσσια πλάσματα ε, που έχουν κέλυφος από ασβέστιο. Λιώνουν τα όστρακα. Δεν έχει ε, υπάρξει ποτέ τόσο όξινο πεχά στον ωκεανό κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. Βλέπετε ε, το ζωοπλανκτόν ας πούμε σε κάποιες εικόνες και αν μειωθεί το πεχά όσο μειωθεί μέχρι το 2050 όπως προβλέπετε τότε αυτά τα μικρά που είναι, ε, πλακτούν που είναι στην ε, αρχή της τροφικής αλυσίδας ε, για την τροφή στον ωκεανό δεν πρόκειται να έχουν την ευκαιρία να αναπτύσσονται καν. Και αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες και οικολογικές για την υδατοκαλλιέργεια και για τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Είδαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τι γίνεται με τους καλλιεργητές στις υδατοκαλλιέργειες που έχουν στρίδια ακριβώς απειλούνται από την οξύνηση των υδάτων. Το ίδιο ισχύει και για το βυθό της Αρκτικής, τα είπε και ο Λίζε, τα θέματα που συνδέονται με τους πάγους. Λοιπόν, να πω το εξής. Όταν μιλούμε για το κόστος της μετάβασης, πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το σχετικό μελλοντικό κόστος. Πλημμύρες, ήδη φέτος το καλοκαίρι Είχαμε άνευ προηγουμένου πλημμύρες, δεν έχουμε ξαναδεί στη Σουηδία τέτοια πράγματα, στις δυτικές ακτές. Είχαμε τεράστιες πυρκαγιές δασικές, τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά όλων των εποχών στη σύγχρονη ιστορία. Στη Σουηδία παρακαλώ. Και αυτό έχει οικονομικό κόστος που θα πρέπει να ε, συζητήσουμε όταν μας απασχολούν τέτοια θέματα και μιλούμε για τις δυσκολίες που έχει η βιομηχανία να κάνει αυτή τη μετάβαση. Επίσης άλλο ενδιαφέρον στο σεμινάριο ήρθε ο πρόεδρος του Euracall, τον, το του Άνθρακα και το ρώτησα εσείς τι κάνετε στη στρατηγική και τα σχέδιά σας για το μέλλον. Πώς προγραμματίζετε, θα σταματήσετε την εξόριξη άνθρακα, γιατί αυτό χρειάζεται, αν θα πρέπει να παραμείνουμε κάτω των δύο βαθμών Κελσίου. Και η απάντηση ήταν ε, όχι, αν είναι δυνατόν, δεν έχουμε καθόλου τέτοια σχέδια να σταματήσουμε τα ανθρακορεχεία. Ενδιαφέρον και αυτό να το γνωρίζουμε. Θα πρέπει να υπάρξουν πραγματικές πολιτικές δεσμεύσεις και σχέδια συγκεκριμένα. Καμιά φορά και απαγορεύσεις. Για να κινηθεί κάπως η βιομηχανία. Και αυτό είναι ευθύνη αυτή τη γενιά, των πολιτικών αυτή τη γενιά. Και θα πρέπει πραγματικά η ενέργεια, η ανανεώσιμη να συμφέρει σε σύγκριση με την ορυκτά κάψιμα. Αυτό δεν ισχύει ακόμα. Φυσικά όσο κοστίζει 5 ευρώ τον τόνο να παράγεις διοξίδιο του άνθρακα να εκπέμπεις προφανώς. Και θα πρέπει η Ευρώπη να είναι φιλόδοξοι με δεσμευτικούς στόχους για τις ανανεώσιμες και την ενεργειακή απόδοση. Ελπίζω να τα καταλάβουμε αυτά, να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων και να λάβουμε αυτές τις τόσο σημαντικές αποφάσεις, ε, το Συμβούλιο δηλαδή, στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τελευταία παρέμβαση. Συνάδελφε Γκριζίπ. Eh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σωστά υπόθηκε ότι ήμασταν υπερβολικά αισιόδοξοι όσον αφορά την Κοπενχάγη. Η αισιοδοξία μας ήταν υπερβολική. Και πολύ συχνά αυτό που συμβαίνει είναι όταν είναι πολύ υψηλές οι προσδοκίες τείνουμε να απογοητευόμαστε ικτρά μετά άμα δεν πραγματοποιούνται. Πολλά έδειχναν ότι η Κοπενχάγη δεν θα ήταν επιτυχία. Ακόμα και σε διμερείς συνομιλίες σαν Πολωνός βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε διμερείς συνομιλίες λάμβαναν τέτοιες πληροφορίες που έδειχναν ότι η σύνοδος κορυφής δεν θα ήταν επιτυχής. Είδαμε ε, ποια ήταν η συμβολή των χωρών με τις περισσότερες εκπομπές και βλέπαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε την επιθυμητή συμφωνία. Απ' την άλλη πλευρά υπήρχαν και κάποια αισιόδοξα μηνύματα όσον αφορά τις συμφωνίες τομεακές της βιομηχανίας για την χρήση των βέλτιστων ε, τεχνολογιών για τη μείωση των εκπομπών. Δεν νομίζω ότι χρησιμοποίησαμε ε, υπόψη μας τις δυνατότητες που υπήρχαν για να βελτιώσουμε τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Θα μπορούσαμε να πετύχει διαφορετικά μεγάλη πρόοδο τα τελευταία πέντε χρόνια. Βήμα-βήμα, αν είχαμε κινηθεί σωστά, θα μπορούσαμε να πετύχει πρόοδο βάσει των βελτίστων διαθεσίμων τεχνολογιών. Είχαν γίνει στη Βαρσοβία κάποιες συναντήσεις στη Τσεχική Δημοκρατία με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών και διαφόρων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της χαλιβουργίας, ε, τσιμεντοπίας κλπ. Λοιπόν έγιναν τέτοιου συναντήσεις. Θέλω να πω το εξή μετά από όλα αυτά. Οι προσδοκίες μου όσον αφορά την επόμενη ε, σύνοδο κορυφής είναι μάλλον μέτριες θα έλεγα ότι τώρα είναι αναπόφευκτο και είναι απόλυτα αναγκαίο να πετύχουμε μια παγκόσμια συμφωνία, εργαζόμαστε υποπίεση, κάτι που θα επιταχύνει την πρόοδο. Δεν θα πετύχουμε τέλειες λύσεις λόγω χρονικής πίεσης, αλλά θα πρέπει να δεχτούμε την πραγματικότητα. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι μπορούμε να έχουμε πολύ καλές προθέσεις, αλλά οι προθέσεις ίσως να αρμηνευτούν διαφορετικά από τους εταίρους μας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η συμφωνία για την μείωση των εκπομπών των αερομεταφορών. Η κατάσταση έχει ως εξής. Κάποιες αεροπορικές εταιρείες δεν παίρνουν χρονοθυρίδες για, να, για υπερπτήσεις πάνω από τη ε, Σιβηρία. Άλλες αγοράζουν τις χρονοθυρίδες. Άλλες που είναι εκτός Ευρώπης αεροπορικές εταιρείες. Άρα γίνονται πιο ανταγωνιστικές αυτές οι εταιρείες εις βάρος του δυναμικού διαχείρισης κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών φορέων ε, που συμμορφώνονται με κάποιους κανόνες. Ας δούμε την ιστορική σκοπιά των πραγμάτων. Η βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετεγκαταστάθηκε μέρη εκτός Ευρώπης λόγω πιο φθηνών εργατικών χεριών, λόγω λιγότερο αυστηρών κανόνων όσον αφορά την παραγωγή. Ε, εδώ και δύο χρόνια είδαμε η τη φαντουργία, κατέρευσε, πάνω από 2.000 άνθρωποι πέθαναν, είχαμε ατύχημα στην Τάκα, στο εργοστάσιο και είδαμε ότι 2.000 κάτοικοι του Μπαγκλαντές εργαζόταν σε αυτό το εργοστάσιο που κατέρευσε ε, για ευρωπαϊκές εταιρείες και πολλούνται τα προϊόντα αυτά στην Ευρώπη και στην Πολωνία μας είχε συγκινήσει η κοινωνική εταιρική ευθύνη, κάτι που είχαμε συζητήσει. Δυστυχώς αρκετές εταιρείες δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές προδιαγραφές και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Οι ντόπιοι υποφέρουν, το κλίμα υποφέρει, το περιβάλλον υποφέρει, αλλά εμείς εποφελούμεθα από όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένα πικρό συμπέρασμα αυτό, αλλά θα πρέπει να το συναγάγουμε σήμερα σε αυτή τη συζήτηση. Ας πω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο κατά τη διάρκεια πολυμερών διαπραγματεύσεων. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη αν θέλουμε να πετύχουμε στόχους που σχετίζονται με την καταπολέμηση αλλαγής του κλίματος. Καμιά φορά η κατάσταση είναι κάπως ε, παράδοξη. Η βιομηχανία η οποία παράγει εξοπλισμό για ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας ανθεί στην Κίνα αιωλική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια κλπ. Αυτός ο τομέας λοιπόν στην Κίνα ανθεί. Όμως η ίδια χώρα εκπέμπει όλο και περισσότερο αέρια του θερμοκηπίου, μολύνει όλο και περισσότερο. Αυτό είναι το παράδοξο. Αυτές λοιπόν οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές, όχι μόνο μεταξύ Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και εντός της Ευρώπης οι διάφορες χώρες έχουν διαφορές. Οι πρόσφατες ε, αποφάσεις που έλαβε η γερμανική κυβέρνηση για περικοπή της στήριξης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έγιναν οι περικοπές όχι διότι δεν χρειάζονται στήριξη παραγωγή ανανεωσίμων πηγών ενέργειας. Μειώθηκε η υποστήριξη διότι επηρέαζε την τιμή της ενέργειας. Η ενέργεια παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίνει να είναι ακριβότερη. Και δεν μπορούν όλα τα κράτη-μέλη να αντέξουν αυτές τις τιμέ. καποια Κάποια κράτη-μέλη αποφασίζουν να ακολουθήσουν διαφορετικό δρόμο, παρόλο που θα ήθελαν να διατηρήσουν τα σχήματα υποστήριξη σε επαρκέ επίπεδο, ούτω ώστε να υπάρχουν ισότιμες συνθήκες στον τομέα και προσπαθώντα να πετύχουμε τους στόχου που έχουμε θέσει. Τέλο, θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά σχετικό με αυτά που κουβεντιάζουμε και τι είναι επανέρχεται όταν κουβεντιάζουμε αυτά τα θέματα. Όταν συζητάμε και για την Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι η γειτονική μας χώρα, έχει αρκετά ενεργοβόρο βιομηχανία, αλλά δεν υπάρχουν μετρήσεις ή υπολογισμοί όσον αφορά τις επιδόσεις των δήμων. Δεν υπάρχουν ε, μονάδες μέτρησης του φυσικού αερίου ένας πρώην υπουργό εξωτερικών, ένας πολιτικός, είπε το εξή σχετικά με αυτό. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία, να τη βοηθήσουμε πραγματικά, ίσως δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε διαφορετικούς δρόμους εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Ίσως θα ήταν καλύτερα να χρηματοδοτήσουμε την αγορά μετρητών φυσικού αερίου. Θα μπορούσε να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό ούτως ώστε να έχουμε κάποια απτά αποτελέσματα, μετρήσεις στα χέρια μας που θα μεταφραζόταν σε αλλαγή προτεραιοτήτων. Προτεραιοτήτων θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν, αλλά θα είχαμε περικοπή κατά 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα περίπου την χρήση ενέργειας στην ε, Ουκρανία. Όταν θέλουμε να ενισχύσουμε την προστασία του κλίματος, μπορούμε να ακολουθήσουμε διάφορες προσεγγίσεις. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση που ταιριάζει σε όλες τις περιστάσεις. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο φιλόδοξους στόχους. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και οι ιδιαιτερότητες. Οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εφόσον θέλει να ηγηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τους γείτονές μας και τους μη Ευρωπαίους εταίρους μας. Ευχαριστώ. Άλλες δύο παρεμβάσεις. Βυσνιεύσκα, συνάδελφε Βυσνιεύσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, χωρίς παγκόσμια συμφωνία για το θέμα του κλίματος, δεν πρόκειται να επιτύχουμε τους στόχους μας. Δεν επιθυμώ να επαναλάβω τα επιχειρήματα που ήδη έχουν αναφέρει άλλο. άλλοι. Έρχομαι μόνο στην παράγραφο 3 του σχεδίου ψηφίσματος. Εδώ και χρόνια Κάνουμε κάθε χρόνο το ίδιο λάθος. Πρόκειται δηλαδή για τις χώρες οι οποίες ήδη έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές τους, δηλαδή στην ουσία οι χώρες μέλη της Ένωσης, οι οποίες ακόμη οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές τους. Βέβαια γνωρίζουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλουμε τις προσπάθειες αυτές. Όμως σημειώστε ότι οι προσπάθειες αυτές είναι ήδη πολύ σημαντικές. Και οι λύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια πρέπει να γίνουν. Πρέπει όμως στις προσπάθειες αυτές να συμμετάσχουν και οι χώρες εκείνες που εκπέμπουν τις μεγαλύτερες ποσότητες αερίων θερμοκηπίου. Εάν αυτές οι χώρες δεν δεσμευτούν να μειώσουν τις εκπομπές τους, δεν θα φτάσουμε ποτέ τους στόχους μας. Να ασκήσουμε μονομερός πίεση για τη μείωση των εκπομπών, αυτό δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει, διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν επιθυμούν να ασκήσουν πίεση στις βιομηχανίες τους για μείωση, μείωση των εκπομπών. Άλλωστε υπάρχει και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός. Ο συνάδελφός μου Ζέμπ μίλησε ήδη για την παραγωγή που λαμβάνει η χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βέβαια υπάρχουν οι κομπές εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη βιομηχανική παραγωγή εκτός που έχει μετακινηθεί προς τις χώρες αυτές όχι μόνο γιατί έχουν φτηνότερα εργατικά χέρια αλλά και διότι οι ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο αυστηρές. Άρα πρέπει, οφείλουμε να διαβουλευτούμε και με αυτούς τους εταίρους, τρίτες χώρες δηλαδή. Έχει απόλυτα ανάγκη των διαπραγματεύσεων αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, τελευταίος αλουχή έσχατος, ο κ. Γκρότε. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα ορισμένες παρεμβάσεις και την τελευταία και όντως δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για το πρόβλημα του κλίματος. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Θα πρέπει να προσέξουμε να παραμείνουμε ρεαλιστές στις παγκόσμιες διασκέψεις και να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Και μέσα στα όρια μας, μέσα στα σύνορά μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε και τι να κάνουμε. να λείπουν τα διδάγματα από εδώ και από εκεί. Είναι πολύ διαφορετικές οι ανάγκες της Πολωνίας από άλλες χώρες της Ευρώπης. Η ανάγκη ασφάλειας της προμήθειας ενέργειας παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο εκεί, πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες χώρες. Μόνο εφόσον συνεργαστούμε στενά μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Και στην Επιτροπή Βιομηχανίας και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουμε βάλει έχουμε καταστρώσει μια πορεία για τη μελλοντική πολιτική του κλίματος. Αν όμως ξεκινήσουμε την προσπάθεια αυτή, πρέπει να γίνει σωστά. Και αν δεν γίνει σωστά, δεν αξίζει το κόπο να γίνει. Τα μεσοβέζικα πράγματα είναι τα χειρότερα. Διότι δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια σχεδιασμού. Κανένας δεν θα αισθάνεται ασφαλής, κανένας δεν θα ξέρει πού βρίσκεται και πού πηγαίνει. Ως θεσμικό όργανο λοιπόν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οφείλουμε να καταστρώσουμε τις συνθήκες πλαίσια και να δεσμευτούμε. Και όχι άλλα να πούμε στο ψήφισμα και αλλιώς να ψηφίσουμε. Στους πανηγυρικούς λόγους που βγάζουν οι πολιτικοί ηγέτες, ωραία λόγια λένε. Όταν όμως έρχεται η ώρα να τα κάνουν πράξη, άρα να επιβαρύνουν διάφορους, δεν τα κάνουν. Εγώ δημοκράτης είμαι. Καμιά φορά θα υπηρεσίσει μια πλευρά, άλλη φορά θα υπηρεσίσει άλλη πλευρά. Όμως, να μην λέμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Άρα, ρεαλιστική προσέγγιση και να δείξουμε ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε, να μην περιμένουμε από τους άλλους. Είμαι απόλυτα πεισμένος για αυτά. Στη Γερμανία έχουμε τις υψηλότερες τιμές ενέργειας. Βλέπω για παράδειγμα ότι στην περιφέρειά μου έχουν σχεδόν καταστραφεί τα ναυπηγεία. Γιατί βρισκόμαστε σε άμεσο ανταγωνισμό με την Νότια Κορέα. Όλες αυτές οι θέσεις απασχόλησης έχουν αντικατασταθεί μόνο από άλλες θέσεις απασχόλησης στις ανανόσιμες ενέργειες που δημιουργεί νέα απασχόληση ο τομέας αυτός. Όλα αυτά σε μια περιφέρεια παράκτια με ασθενείς διαθρώσεις, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλή η, ε, είναι πολύ ψηλός ο διεθνής ανταγωνισμός. Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να αποσυνδεθεί από τις εκπομπές των διοξιδιών του άνθρακα. Αυτή πρέπει να είναι η εξέλιξη. Οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να έχουν δουλειά, να βγάζουν το ψωμί τους. Δεν υπάρχει ούτε για τη Γερμανία, ούτε για την Πολωνία, ούτε για την Κύπρο, την Ισπανία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δεν υπάρχει καμιά μαγική συνταγή. Άμα θέλετε να μιλήσετε για ατομική ενέργεια, μην έρθετε να μιλήσετε στους Γερμανούς Σοσιαλδημοκράτες. Με τους Γάλλους μπορείτε να μιλήσετε όμως. Ας δούμε καλύτερα λοιπόν ποια πράγματα μας ενώνουν, ποια πράγματα εξασφαλίζουν μια συνοχή και να συνεχίσουμε μια πορεία, να, να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε μια πορεία, αλλά με συνέπεια. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για αυτή τη συζήτηση, την πλουσιότατη. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επίτροπη, την κυρία Μπάρντραμ, για την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα στα αξιότιμα μέλη. Ξεκινώ ευχαριστώντας το Κοινοβούλιο για την εμπεριστατωμένη αυτή συζήτηση που δείχνει τον πλούτο και το βάθος. Η ενδελέχεια της συζητήσεως δείχνει ότι υπάρχει η κατανόηση των διακυβευμάτων και το μέγεθος των προκλήσεων είναι επίσης γνωστό που έχουν μπροστά μας. Το παγκόσμιο πλαίσιο υπόσχεται πολλά σήμερα. Φαίνεται αρκετά θετικό. Το Σαββατοκύριακο μου στη Νέα Υόρκη είδα τις εκατοντάδες χιλιάδες των ανθρώπων στους δρόμους. Άκουσα πολλούς ηγέτες να ομιλούν όχι μόνο στη Σύνοδο Κορυφή, αλλά και σε συνδυάσει του Φόρουμ της Μεγάλης Οικονομίας για τις υποχρεώσεις που έπρεπε να αναλυφθούν, την προθυμία που υπάρχει να συμμετάσχουν σε συλλογικέ παγκόσμιες προσπάθειε. Οι βασικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ενώσης κινούνται. Κυρίως η δράση για το κλίμα στις ΗΠΑ είναι άνευ προηγουμένου. Πολλά επιτυγχάνονται μέσω διαφόρων εκτελεστικών διαταγμάτων και εντολών, αλλά οι δραστηριότητες της ΣΥΠΑ ε, φτάνουν σε διαφορετικό επίπεδο. Και η Κίνα κινείται. Έχει το 12ο πενταετές ε, σχέδιο και εμπεριέχει περιβαλλοντικές στοιχεία. Συνεργαζόμαστε με τους Κινέζους, εταίρους μας, όσον αφορά το όλο σχήμα και το πρόγραμμα ανταλλαγής ρήπων που θα εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο. Βλέποντας τις παλαιότερες πολιτικές που ακολουθήσαμε, είναι σημαντικό ότι η αποσύνδεση ανάπτυξης από την αύξηση των εκπομπών είναι κάτι που παρατηρήσαμε και παρατηρούν και οι εταίροι μας. Έχουμε εφαρμόσει πιο περίπλοκες νομοθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι κάτι που ενδιαφέρει τους εταίρους μας αυτό. Θέλουν και αυτοί έχουν την προσδοκία να κάνουν παρόμοια βήματα για μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ένα από τα παραδείγματα της στήριξης αυτής είναι στη σύνοδο κορφής του Ban Ki-moon, υποστήριξη από την Παγκόσμια Τράπεζα όσον αφορά την τιμή του άνθρακα. 73 χώρες και διάφοροι περιφερειακοί οργανισμοί και πάνω από χίλιες εταιρείε υποστήριξαν τη δήλωση της Παγκόσμιας Τράπεζας και δείχνει αλλαγή του ρεύματος. Παραδέχονται ότι κοστίζει η έλλειψη δράσης και θέλουν να δώσουν κίνητρα για δράση. Πρέπει να συνεχίσουμε στο μονοπάτι το φιλόδοξο. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του IPCC, του Διακυβερνητικού Πάνελ για την Αλλαγή του Κλίματος, χωρίς δράση που έχει νόημα και χωρίς συμφωνία στο Παρίσι, με μεγάλη συμμετοχή, ο μέσος όρος αύξηση δημοκρασίας μπορεί να φτάσει 3,5 μέχρι 4 βαθμούς μάλλον αύξηση Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα. Το έχουν παραδεχτεί και άλλοι εταίροι ότι υπάρχει αυτός ο σχετισμός, μπαίνουμε σε κρίσιμη φάση. Η διάσκεψη της Λίμα πρέπει να δώσει αποφάσεις και συμφωνίες που θα μας επιτρέψουν να ακολουθήσουμε συγκεκριμένες διαδικασίες εν ώψη Παρισιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θέλει. Να καθορίσει τις απαιτήσει για πληροφορίες. Πληροφορίες που θα ενημερώνει τους εταίρους και πώς μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση διοξιδίου του άνθρακος, εκπομπών διοξιδίου του Να κάνουν σωστή αξιολόγηση. Να δουν τα μέτρα που εφαρμόζονται είναι τα σωστά και δίκαια. Θέλουμε να έχουμε γενική εικόνα, πραγματική εικόνα για το που βρισκόμαστε. Σαν παγκόσμια κοινότητα για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο της αύξησης θερμοκρασίας κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η πορεία της διεθνούς κοινότητας στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου. Πρέπει να εξασφαλίσουμε και κάτι άλλο. Η Συμφωνία των Παρισίων να είναι βιώσιμη μακροχρόνια αν υπάρχει μεταξύ, διαφορά μεταξύ των δύο βαθμών και των παγκόσμιων φιλοδοξιών, υπάρχει μηχανισμός να επανέλθουν τα μέρη προς αναθεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη τεχνολογίας εξελίξεις. Τι λέει η επιστήμη. Και να αυξήσουν ανάλογα τις φιλοδοξίες τους. Χρειάζεται να συμπορευτούμε με την ε, επιστήμη και τα επιστημονικά απορίσματα της ανακαλύψης. Πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε τη σωστή προσαρμογή, να καλύψουν τι οικονομικέ ανάγκε των αναπτυσσομένων χωρών. Χαίρομαι που το σχέδιο ψηφίσματό σα το τονίζει. Το πώ βλέπουν τα πράγματα οι αναπτυγμένε χώρε χρειάζεται επεξεργασία. Πρέπει να έχουμε διαδικασία που είναι πραγματική και πιστευτή για του εταίρου μα, Να αισθάνονται ότι μπορούν να συμμετάσχουν οι εταίροι μα στην όλη προσπάθεια. Να καταπολεμήσουν την αλλαγή του κλίματο αλλά και να μπορέσουν να προσαρμοστούν δεόντω. Τέλος. Στη Λίμα τι πρέπει να πετύχουμε. Να έχουμε ένα σχέδιο κειμένου με τα βασικά στοιχεία. Απομένουν 14 μήνες για το Παρίσι. Πρέπει το κείμενο για την επαγμάτευση να είναι επιτάπητος, να είναι έγκαιρα διαθέσιμο πριν τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις των Παρισίων. Στη Λίμα ήδη πρέπει να έχουμε καλή εικόνα να βλέπουμε τα κομμάτια του παζλ και να πετύχουμε ένα πακέτο πολιτικά ισορροπημένο που μπορεί να καλύψει όλες τις χώρες και να επιτρέπει συλλογική προσπάθεια. Και έτσι τελικά μπορούμε να ακολουθήσουμε το μονοπάτι που θα μας οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου της ε, αύξησης θερμοκρασίας κατά λιγότερο από δύο βαθμούς σε μέσο όρο στον κόσμο. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος. Πιστεύω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε έτσι εδώ τη συζήτηση από το συγκεκριμένο σημείο. Το μόνο που απομένει είναι το χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα προθεσμίες τροπολογίες για το ψήφισμα 8 Οκτωβρίου στις 12 ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΝΒΗ 5 Νοεμβρίου και μετά ψηφίσουμε στην Ολομέλεια 24 Νοεμβρίου στη Σύνοδό μας στο Στρασβούργο. Εξαντλήσαμε λοιπόν και το σημείο 17, όπως σας είχα πει στην αρχή, αλλάξαμε την ημερήσια διάταξη προσθέτοντας ένα σημείο αφορούσε αυτό προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποια χαρτοφυλάκια που αφορούν το περιβάλλον, κάποιες υποθέσεις του περιβάλλοντος οι πράσινοι το ζήτησαν αυτό. Ο Σάιφος Ικάουτ θα δώσω λοιπόν το λόγο στον συνάδελφο για να μας παρουσιάσει το όλο θέμα και μετά το λόγο θα έχει η Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Συνάδελφοι Ικάουτ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι το τελευταίο και μετά δεν θα ξαναμιλήσω, σας το υπόσχομαι. Για σήμερα. Είναι μια συνέχεια που δίνουμε στην επίσκεψη του Επιτρόπου Ποτότσνικ στην Επιτροπή μας εδώ, έμβη, πριν τις έννοιες διακοπές, όπου ξεκαθάρισε ο Επίτροπος ότι αν δείτε τις προτάσεις που αναφέρουμε στην προφορική ερώτηση που είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, ε, βιώσιμη κατανάλωση τροφίμων και ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές, ουσιαστικά μας είπε ότι είναι έτοιμο το υλικό να φύγει. Ωστόσο, δεν έχουμε δει τίποτα από αυτές τις προτάσεις ακόμα. Και λίγο μας προβληματίζει τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι γίνεται εκεί πέρα, διότι ταυτόχρονα Όλες αυτές οι προτάσεις είχαν αναφερθεί στο πρόγραμμα εργασίας. Δηλαδή κάπου είναι κοινοποιημένε, κάπου τους έχουν ανακοινώσει ότι επίκυνται. Εμείς ως Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχουμε κάνει είτε ψηφίσματα είτε εκθέσεις πρωτοβουλίας. Επ' αυτού είναι όλα έτοιμα λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η υπόθεση και παρόλα αυτά κάπου έχει μπλεχτεί και μας προβληματίζει μας πρασίνουσε εκεί τι τρέχει. Τι εμποδίζει επιτέλους την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τις προτάσεις της. Και ακόμα πιο σημαντικό για μας είναι να δείτε, αν διαβάσετε το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, που είναι νομοθετικά δεσμευτικό, είναι ευρωπαϊκός νόμος. Και να σας παραθέσω μερικά στοιχεία. Για παράδειγμα, μία από τις προϊότητες, στόχος 4, οι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει, θα έχουν ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Δηλαδή, πιο σαφής πεθαίνεις. Ε, ε, επίσης, στο ίδιο στόχο 4, Ευρωπαϊκή Ένωση θα επεκτείνει ε, τις απαιτήσεις για τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις και θα έχει δεσμευτικά κριτήρια. Δηλαδή είναι νόμος όλα αυτά, γιατί δεν εφαρμόζεται. Αν δείτε για τις ουσίες που προκαλούν εδώ κλινικές διαταραχές, το ίδιο πρόγραμμα λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, αντιμετωπίσει το θέμα σε όλη την κοινοτική νομοθεσία, τη σχετική. Δηλαδή, όχι μόνο ακούσαμε από τον Επίτροπο Ποτότσνικ ότι είναι έτοιμα να ξεκινήσουν όλα αυτά, όχι μόνο το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα να προχωρήσει, όχι μόνο το αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα ε, δράση τη. αλλά στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον που είναι νομοθετικού περιεχομένου και έχουν συναποφασίσει κοινοβούλιο και συμβούλιο. Ερώτηση. Γιατί ολιγορείτε. Και ποιον δεν δεσμεύει από ό,τι φαίνεται το 7ο πλαίσιο για το περιβάλλον. Αυτή είναι η ερώτηση προς την Κομισιόν. Γιατί όλοι ξέρουμε ποιος μπλοκάρει. Είναι σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν μετά τη σημερινή συζήτηση δεν μπορεί κανείς να μας υποσχεθεί και να δεσμευτεί ότι θα φέρει αυτά τα θέματα, μήπως την άλλη φορά να καλέσουμε το Γενικό Γραμματέα στην ΕΜΒΗ για να μας απαντήσει. Γιατί υποθέτω ότι και ο Γενικός Γραμματέας δεσμεύεται από το 7ο ή Γενική Γραμματέας. Εάν δεν δεσμεύεται, να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί εκεί θα έχει ενδιαφέρον πια η συζήτηση. Ξέρω ότι θέλουν όλοι οι συνάδελφοι να μιλήσουν για ε, τα πιο ειδικά ζητήματα. Αυτή είναι η γενικότερη ερώτηση. Να μας την απαντήσετε και μετά θα κάνουμε και τις επιμέρους ερωτήσεις μάλλον. Εγώ θα ήθελα να δώσω αμέσως το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μία πρώτη ανάλυση του θέματος σε σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφος Ριχάουτ. Μετά θα έχουμε παρεμβάσει των άλλων συναδέλφων που ίσως θέλουν να θέσουν κάποιες ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα δώσουμε το λόγο στο τέλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very much, uh, Mr. Uh, President. And... Ευχαριστώ και καλό σας απόγευμα. Προσκαλέσατε σήμερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στην προφορική αυτή ερώτηση σε συνέχεια της πολιτικής παρεμβάσεως του Επιτρόπου Ποτότσνικ που έλαβε χώρα εδώ ενώπιον σας αρχές Σεπτεμβρίου. Πρώτα θα σας επιβεβαιώσω ότι η οι υπηρεσίες της Επιτροπές ακολουθούν τις γραμμές του 7ου προγράμματος όπως εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πέρσι τον Οκτώβριο μετά από πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακολουθούμε τις γραμμές του 7ου προγράμματος δράσεως όχι μόνο σε γενικές γραμμές αλλά και στη λεπτομέρεια αναφορικά με τις διάφορες πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται εκεί Έχουμε δώσει τη σχετική συνέχεια με τα απαραίτητα προπαρασκευαστικά μέτρα, αλλά και με εργασία επί της ουσίας. Και για τις τέσσερις αυτές προτάσεις. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη, περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, γι' αυτά σας επιβεβαιώνω ότι οι υπηρεσίες μας έχουν συντάξει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες καθώς και την μελέτη αντικτύπου που απαιτείται διαδικαστικά Δύο λοιπόν αντίκτυποι μελέτης που έχουν ελεγχθεί και από το Impact Assessment Board της Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα, τα απορρίμματα τροφίμων, ίσως να τα γνωρίζετε καλύτερα και τα πράγματα γιατί ήταν κάπως πιο ορατή η δράση της Κομισιόν, η οποία Κομισιόν ενέκρινε πριν από το καλοκαίρι φέτος δέσμη μέτρων για την αναθεώρηση της πολιτικής και των στόχων για τα απορρίμματα συντάχθηκε ανακοίνωση από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το λεγόμενο αγγλιστή food waste που όμως τελικά δεν αποτέλεσε μέρος της δέσμης που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρόλα αυτά εφιστώ την προσοχή σας σε ένα σημαντικό θέμα την υποχρέωση δηλαδή καλύτερης μέτρησης των επιπέδων του food waste και των άλλων σχετικών και τον μη δεσμευτικό στόχο της μείωσης του food waste κατά 30% μέχρι το 2025. Αυτά έχουν περιληφθεί στην νομοθετική πρόταση. Άλλα στοιχεία συνεχίζουν να εξετάζονται από τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλα στοιχεία δεν έχουν περιληφθεί στην πρόταση που ενεκρίθη πριν από το καλοκαίρι. Αναφορικά τώρα με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, επιβεβαιώνω επίσης ότι η σχετική προπαρασκευαστική εργασία μεταξύ αυτής και οι επιστημονικές εμπειρογνωμοσύνες και η συλλογή των δεδομένων έχουν ήδη εξαχθεί από τις υπηρεσίες της Κομισιόν και κάποια στιγμή μάλιστα το προπαρασκευαστικό αυτό έργο ξέφυγε από τα όρια λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε και την συμβολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ασφάλειας τροφίμων του Κοινού Κέντρου Ερευνών που συνέβαλαν με δεδομένα που είναι απαραίτητα για την θέσπιση των επιστημονικών πτυχών για τα κριτήρια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε γενικές γραμμές έχει ολοκληρωθεί το έργο, προπαρασκευής του ουσιώδους περιεχόμενου της προτάσεως. Βέβαια, σημειώνω ότι τουλάχιστον ορισμένες από τις τέσσερις προτάσεις δεν περιελήφθησαν επισήμως στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τουλάχιστον για το 2014. Τουλάχιστον όχι στο πρώτο τμήμα του προγράμματος εργασιών που θεωρεί η Κομισιόν ότι είναι δεσμευτικό. Αυτό πάλι με τη σειρά του σημαίνει ότι για την έγκριση πρωτοβουλίας απαιτούνται δύο στοιχεία. Η τεχνική προπαρασκευή και η πολιτική απόφαση. Η τεχνική προπαρασκευή λοιπόν λίγο πολύ έχει ολοκληρωθεί. Το περιεχόμενο των προτάσεων είναι έτοιμο η πολιτική απόφαση μένει να ληφθεί έτσι ώστε να προχωρήσουν οι προτάσεις αυτές. Δεν θα είναι ρεαλιστικό βέβαια να πει κανείς ότι η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί στους τελευταίους μήνες ή εβδομάδες της λειτουργίας του Συλλογικού Σώματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που η θητεία της λύγει, αλλά πάντως το μέγα μέρος της προπαρασκευαστικής εργασίας έχει γίνει για λογαριασμό και της μελλοντική Επιτροπής. Και η δική σας Επιτροπή θα έχει το χρόνο να εξετάσει σε βάθος. Να εξετάσετε δηλαδή κι εσείς τις τέσσερις πρωτοβουλίες, να κρίνετε και να κρίνουμε και εμείς για το περιεχόμενο και για το αν τελικώς θα εγκριθούν ή όχι και εάν εγκριθούν, πώς. Αυτή είναι η δική μου παρέμβαση. Είμαι βεβαίως στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Στον βαθμό βέβαια που μπορώ να απαντήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αφού ήρθαμε εδώ, ας ακούσουμε τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Συνάδελφε Στάες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα επικεντρωθώ στα τρόφιμα εγώ, στο συγκεκριμένο φάκελο, στην παρέμβασή μου, με εκπλήσει αυτά που έρχεται εδώ να μας διηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2013, δηλαδή έχει περάσει λίγος χρόνος, ανήγγειλε ότι θα φέρει ανακοίνωση για τη βιώσιμη πολιτική για τα τρόφιμα, που είναι περισσότερο από τη σπατάλη τροφίμων, δεν είναι μόνο food waste, ε, είναι πολύ ευρύτερο. Τον Απρίλιο του 2013 το είπε και γύρω στα τέλη του 2013 και αρχές του 2014 πρόκειτο να το φέρει. Ο Επίτροπος Ποτόσνικ εδώ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή επανειλημμένα δήλωσε ότι είχε περίπου ολοκληρωθεί η δουλειά αυτή και παραμονές των εκλογών άφησε να εννοηθεί ότι θα ανακοινωνόταν και θα εγκρινόταν αυτή η ανακοίνωση από το Σώμα των Επιτρόπων δηλαδή στη συνεδρίαση της 7ης Μαΐου, δυόμιση εβδομάδες πριν τις εκλογές κατόπιν πιέσεως, από ό,τι καταλαβαίνω, της Γενικής Γραμματέως και του ίδιου του Προέδρου Μπαρόσο, βγήκε από την ημερήσια διάταξη ε, για να μην επηρεάσει, λέει, φοβόντουσαν την προεκλογική εκστρατεία και είπαν ότι η ανακοίνωση θα έρθει μην ανισχύεται αμέσω μετά τις εκλογές. Ε, όντως, ε, μετά τις εκλογές μιλήσανε για την κυκλική οικονομία όπου υπάρχουν διάφορα πράγματα για τη σπατάλη των φήμων και το θέμα αυτό, αλλά ως ανακοίνωση αυτή καθ' αυτή δεν ήρθε. Και περιμένουμε τώρα, εννιά μήνες μετά βράζουμε στο ζουμί μας και η ε, δικαιολογία είναι ότι σε λίγες ομάδες αναλαμβάνει η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε θα αρχίσουμε από την αρχή. Μα είναι πολύ καλό το κείμενο που έχει ήδη ε, γραφεία από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν επενδύσει σε αυτό. Έχει γίνει δημόσια διαβούλευση, ψήφισμα του Κοινοβουλίου το 2012 παρακαλώ. Οπότε όλα είναι έτοιμα. Στο μεταξύ έχει διαρρεύσει και το κείμενο και θέλω να συγχαρώ τους συντάκτες και τον Επίτροπο Ποτότσνη κυκλοφορεί στον τύπο. Και δεν μπορώ να καταλάβω και υπό το φως των συζητήσεων που είχαμε εδώ για παράδειγμα για την εκπομπή ε, αερίων του θερμοκηπίου και όλα αυτά για το κλίμα, το, το κλίμα που συζητούμε, ότι δεν τολμάει η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα καλό έγγραφο να το φέρει στη δημόσια συζήτηση, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε επιτέλους αυτή τη συζήτηση. Αφήστε δε που για μένα είναι και ε, ντροπή που δεν έχει συμπεριληφθεί αυτό σε μια γενικότερα νομοθετική πρωτοβουλία. Ερωτώ. Υπάρχουν άλλες εξουσίες πάνω από τον κύριο Ποτότσινγκ, πάνω από τον Επίτροπο Τσόλος, πάνω από τον Επίτροπο ε, που είναι αρμόδιος για ζητήματα, πώς το της κλιματικής αλλαγής. Ποιος έχει βάλει το χέρι του εκεί και έχει σταματήσει αυτό. Ο ίδιος ο κύριος Μπαρόσο και η κυρία Ντέι ε, είναι τροχοπέδη σε αυτή την υπόθεση. Παρακαλώ να μου το επιβεβαιώσετε. Και συμφωνώ με τον Μπάς Εκχάουτ, αν δεν μας απαντήσετε θα καλέσουμε την κυρία Ντέι ή τον ίδιο τον κύριο Μπαρόσο να μας τα εξηγήσει λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ. Αντιπρόεδρε Τζάβορ, έχετε το λόγο. Mr. President, dear colleague. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφε και εγώ, όπως και ο Σταές, θα ήθελα να θέσω το θέμα των περιβαλλοντικών ελέγχων. Αυτοί έχουν κρίσιμο ρόλο να παίξουν. Εξασφαλίζεται έτσι η ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το περιβάλλον. Σημαντικότατο ζήτημα. Ακόμα και το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη ζήτησε νομοθετική πρόταση μέχρι το τέλος του 2009. Τώρα έχουμε τέλος 2014 και τίποτα δεν έχει προταθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι απαράδεκτο κατά την άποψή μου. Είναι μεγάλο εμπόδιο όσον αφορά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου. Ερώτηση βάσει τον όποιο ο Στάρες. Γιατί αυτή η πρόταση δεν ήρθε. Μας είπαν ότι ήταν ε, αρχές του έτους έτοιμη. Έχει γίνει εξολόγηση αντιχτύπου. Υπήρξε θετική τοποθέτηση του, Συμβουλίου για την εξολόγηση των ε, συνεπειών. Έγινε η ε, ανάλυση. Γιατί δεν έχει υποβληθεί πρόταση από τις αρχές του καλοκαιριού. Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη τώρα αφορά τους περιβολοντικούς ελέγχους, διότι το θέμα των ε, απορριμμάτων από τρόφιμα ε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν αναφέρεται καν ο περιβαλλοντικός έλεγχος. Σε καμία ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κανένα έγγραφο. Ερώτηση. Ξανά. Ποιος μπλοκάρει την πρόταση. Γιατί δεν μας έχει υποβληθεί. Τι εγγύηση έχουμε ότι η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει σε μια ταχεία έγκριση, υιοθέτηση αυτού, αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ. Γκερμπράντι για τους φιλελεύθερους. Συγγνώμη Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους πράσινους που έθεσαν το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη. Βέβαια ο χρονισμός είναι κάπως ατυχής. Τέλος πάντων, ετέθη. Πριν από δύο χρόνια ανέλαβα μια πρωτοβουλία. Ετοίμασα μια επιστολή εκ μέρους Επιτροπής Περιβάλλοντος. Απευθυνόμαστε στον πρόεδρο Μπαρόσο και διαμαρτυρήθηκε για το ίδιο θέμα. Ε, είναι στο λέγεται σαν τάφος, ένα σιρτάρι που έχει θάψει πολλές προτάσεις. Έτοιμες οι προτάσεις να δημοσιευθούν. Στο σιρτάρι της κυρίας Ντέι έχουν θαυτεί. Βλέπω ότι κάποιοι εξωματούχοι χαμογελούν. Νομίζω ότι κάποιο νεύρο έχω ακουμπήσει. Κάπως δεν πέρασαν λοιπόν οι προτάσεις από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα. Βλέποντας λοιπόν το νέο πρόγραμμα της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτά που υπόσχονται οι υποψήφοι επίτροποι, αυτό το σιρτάρι τώρα του Γενικού Γραμματέα έχει βγει έξω από τον παρελαιμόν πλέον. Είναι η μαύρη τρύπα. Η μαύρη τρύπα ήταν πριν ένα σιρτάρι και τώρα έχει το μέγεθος σχεδόν ε, το, όσο το μισό μπαρλεμού. Πολιτικός πως αυτό είναι απαράδεκτο. Εάν σε ένα εθνικό κοινοβούλιο, αν ένας υπουργό υπόσχεται κάτι και δεν τη τηρήσει, θα τον ε, διώξει το κοινοβούλιο. Κάπως αυτό το κοινοβούλιο τα πράγματα πάνε διαφορετικά. Δεν καταλαβαίνω. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέρνει και ξεφεύγει έτσι. Εντάξει, είμαστε στην τελευταία φάση, τελική φάση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της δεύτερη του κυρίου Μπαρόζο και δεν περιμένω καμία άλλη πρόταση πλέον αλλά πιστεύω ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου πει και παραθέτω να ακολουθήσει το 7ο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσεως λεπτομερώς, φαντάζομαι ότι αυτό το πρόγραμμα δράσης το 7ο μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα του περιβάλλοντος. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μια πολιτική υπόσχεση και της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, κάθε υπόσχεση που δίδεται όσον αφορά το 7ο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσεως που δεν το υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι και ένας λόγος να ζητήσουμε από τον Πρόεδρο Γιούνκερ να έρθει στην Ολομέλεια στην Επιτροπή μας. Αν περί αυτού πρόκειται, είμαστε ακόμα στην αρχή μιας τεράστιας ε, πολιτικής διαμάχης. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Άουκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι στα όσα λέχθηκαν. Ήμουν 20 χρόνια στο Δανέζικο Κοινοβούλιο. Τα ίδια πράγματα πέρασαν μέσα από την νομοθετική διαδικασία και είναι νόμος. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε πολιτική επιβεβαιώση των όσων έχουμε ήδη εγκρίνει. Το πρόγραμμα δράσεων Έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης, είχε έρθει το Συμβούλιο, όλοι ήταν εκεί και ψηφίστηκε. Και όχι υπογείως, με πραγματικές πολιτικές αποφάσεις. Το χρειαζόμαστε λοιπόν αυτό και αυτό πραγματικά με ανησυχεί, γιατί υπάρχουν βέβαια διάφορες υποθέσεις, αλλά το πρόγραμμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη είναι το δικό μας μωρό, δανέζικο και της δικής μας πολιτικής οικογένειας. Είμαστε πολύ περήφανες, διότι το εφαρμόσαμε σε όλες τις χώρες μέλη. Γιατί δίνει στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αυτή την πρόσβαση. Λοιπόν αυτό έγινε και μετά σταμάτησε εδώ στην Ένωση. Είχαμε πει ότι αν τροποποιηθεί θα το εγκρίνουμε τελικά. Δίνει το δικαίωμα στους πολίτες. Και είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό για να ενισχύσουμε την αξιοπιστία του Ευρωκοινοβουλίου και του συστήματος. Και είναι πολύ ανησυχητικό που βλέπουμε η νέα Κομισιόν να προσπαθεί να μειώσει την αξία του. Τώρα για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Στη χώρα μου τουλάχιστον, την Δανία, αλλά νομίζω και σε άλλες πολλές, αυτό μπήκε και στην προεκλογική εκστρατεία, διότι πριν από τις εκλογές είχε παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Εμείς μπορέσαμε να αποδείξουμε την επιρροή που έχει στα έμβρια, στα αγέννητα παιδιά και στην ανδρική γονιμότητα. Ήμουν σίγουροι ότι όλοι θα κατέβουν στις διαδηλώσεις αν δουν ότι αυτά τα πράγματα μειώνουν τη γονιμότητά τους. Και βλέπουμε τώρα υπάρχει και η μελέτη. Και όμως δεν συμβαίνει τίποτε. Εμείς υποσχεθήκαμε στην προεκλογική εκστρατεία ότι το θέμα υπήρχε και μας το είχαν υποσχεθεί ότι θα προχωρήσει. Νομίζω ότι από το 98 χρονολογείται ο προηγούμενος κανονισμός. Έχει κινητοποιηθεί τώρα. Εμείς θα χρειαστεί να κινητοποιηθούμε με τη σειρά μας. Και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν χρειάζεται να κινητοποιηθούμε κατά της Κομισιόν. Μπορούμε να το προχωρήσουμε αφού θέλουμε να διαθέτουμε πολιτική αξιοπιστία. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να πείτε όχι μόνο στον Ποτότσνικ, αλλά και σε αυτό το Ιρλανδικό φάντασμα που έχουμε ακούσει τόσο πολλές φορές, γιατί η Ιρλανδική Προεδρία ζήτησε την εφαρμογή του και την τελικοποίησή του, του προγράμματος δράσεων δηλαδή. Αναμένω την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Έχουμε τελευταία παρέμβαση του συνάδελφου Τόρβαλτς. Δεν έχουν ζητήσει άλλοι το λόγο και μετά δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορίστε. Σύντομα. Σύντομα. Ε, ε, ήταν αστείο έτσι με θλιβερό τρόπο να ακούμε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύντομα. Ε, να το πω ότι όλα έχουν γίνει αλλά δεν συνέβη τίποτα που μου θυμίζει ε, μια ιστορία στη δεκαετία του 30 από ένα ρωσικό κολχός. Ε, σύντροφε Στάλιν, κάναμε τα πάντα, αλλά δεν έχει μαζευτεί σοδιά. E Ευχαριστώ. Το λόγο τον έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα ήθελα να απαντήσω γενικώς αναφερόμενος στις στοιχείες στις οποίες μπορώ να απαντήσω. Θέλω να πω ότι αν πέρασε ο χρόνος προσπαθήσαμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά ενισχύοντας το όλο έργο και την επιστημονική διάσταση τις πληροφορίες τα επιχειρήματα, συνεργαζόμενοι με επιστήμονες, συνεργαζόμενοι με δίκτυα επαγγελματιών, επιθεωρητές του τομέα του περιβάλλοντος και με άλλους επαγγελματίες, ούτως ώστε να αυξήσουμε την αποδοχή των ιδεών που αποτελούν τη βάση των προθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεργαστήκαμε και με τα κράτη-μέλη και εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε με αυτά προς διευκόλυνση της αποδοχής των ιδεών και προς διευκόλυνση της διαδρομής των προτάσεων από τη στιγμή που θα εθετηθούν. Τελικό σχόλιο. Κάποιος βουλευτής αναφέρθηκε σε αυτό. Το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα, θεμητό αυτό, δικαιολογείται και από τις πραγματικές εξελίξεις στον κόσμο. Εάν εθελοτυφλούμε όσον αφορά τις εξελίξεις, και να μην δεχόμαστε ότι χρειάζεται δράση θα ήταν κάτι μη ορθό. Φρονούμε ότι ότι είναι θεμητό το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για αυτά τα θέματα, πρέπει να συνεχιστεί και εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το διάλογο, τον ουσιαστικό με το Κοινοβούλιο για όλα αυτά. Αν συνεχίσει το Κοινοβούλιο να στηρίζει τη δράση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά τα θέματα, θα εισακουστεί το πολιτικό μήνυμα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντηση. Και εδώ με το πρόσθετο σημείο της ημερήσιας διάταξης ολοκληρώνουμε τη συνεδρίαση την απογευματινή. Αύριο το πρωί θα ξαναρχίσουμε στις 10 μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών. Καλό σας βράδυ.